δεν, μπορώ δεν πρέπει να διαμαρτυρηθούμε μόνο για την απουσία του Συμβουλίου. Λείπει και ο Γενικό Γραμματέα του ίδιου του Κοινοβουλίου. Ενώ έχουμε να του πούμε διάφορα για το Κοινοβούλιο. Θα έπρεπε και αυτό να είναι εδώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Γενικό Γραμματέας σίγουρα θα έρθει λίγο αργότερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Ας αρχίσουμε τη συζήτηση. Πρώτο είναι ο Γιάννη Κάια, ο εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σα, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε και κύριοι. Θα ήθελα από το σημείο αυτό να πω ότι είναι σχετικά δύσκολη η διαδικασία κατά την άποψή μου να αρχίζει κανείς μια συζήτηση χωρίς να είναι παρόντες αυτοί ε, που θα πρέπει να τους δώσουμε την απαλλαγή και θα πρέπει να συζητήσουμε ε, για το ε, εάν και κατά πόσο θα αναβάλουμε την απαλλαγή, θα τη δώσουμε ή όχι. Εγώ γνωρίζω πολλούς συναδέλφους ε, που είναι παρόντες από την Επιτροπή. Ξέρουμε και τις θέσεις μας ο καθένας. Καλό είναι να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων και φιλικό, αλλά χρήσιμο δεν είναι. Γι' αυτό θα πρότεινα να το συζητήσει η Επιτροπή Ελέγχου να ε, καλούμε επίσημα τα όργανα περί των οποίων πρόκειται στην απαλλαγή και αν δεν είναι παρόντα να αναβάλουμε τη συζήτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία. Χρηματοπιστωτική κρίση έχει ως συνέπεια ε, να ελέγχουν ε, όλες οι κυβερνήσεις τους προπολογισμού και ε, κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν. Είμαστε στο πρώτο έτος μιας νέας θητείας του Κοινοβουλίου, έχουμε και νέα επιτροπή και τώρα συζητάμε ε, την απαλλαγή του 2008 της παλιάς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλές νέες προοπτικές τώρα. Χρειάζεται νέα νοοτροπία και νέα αντιμετώπιση από τα κράτη-μέλη. Γιατί για πρώτη φορά ε, τους ορίζει συνυπεύθυνους ε, η συνθήκη της για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στην απαλλαγή του 2008 θέλησε ο εισηγητής να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί στη ε, βελτίωση του ελέγχου του προπολογισμού και ε, μαζί με αυτή τα κράτη-μέλη. Η ομάδα μας στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θέλει ε, κάθε χρόνο βελτιώνονται οι εκθέσεις για την απαλλαγή και με τη βοήθεια του ελεγκτικού συνεδρίου. Το Συμβούλιο έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο κλειδί ω προ τα κράτη-μέλη και καλό θα ήταν και χρήσιμο να μα βοηθήσει και το ελεγκτικό συνέδριο για να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα που έχουμε, ο προπολογισμό έχει αιτήσιο χαρακτήρα. Πολλά προγράμματα τη Ένωση έχουν πολιετή χαρακτήρα. Και ανησυχούμε ιδιαίτερα σε κάποιου τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εφαρμόσει τι προτεραιότητε τη. Παραδείγματα. Συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό τα ε, χρήματα και τα κονδύλια που δίνονται στα διαρθρωτικά ταμεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εδώ θα πρέπει να έχουμε απλούς κανόνες και ε, επιστροφή ε, αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Το ελεκτικό συνέδριο μπορεί να μας ε, βοηθήσει να εντοπίσουμε καλύτερα τις ατασταλίες. Γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα δράσης για τα τα μία προβλέπει την ανάκτηση των πόρων. Αναμένουμε την εξέλιξη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ταμεία προβλέπει την ανάκτηση των πόρων. Αναμένουμε την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας. Υπάρχει μια διαδικασία επίσης προενταξιακή στις υποψήφιες χώρες για να ε, τις βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Αλλά δεν θα πρέπει να τορπιλίζεται ο στόχος από παραθυράκια. Γι' αυτό παρακαλώ να απορρίψετε τις τροπολογίες του ΕΛΚ που ε, ε, κάνει κάποιες προτάσεις για την Τουρκία, για την προταξιακή βοήθεια. Ε, θα πρέπει να διοριστεί νέος διευθυντής στην Όλαφ, φωτογραφή πολέμηση της απάτης για να τελειώνει αυτή η συζήτηση και να υλοποιηθούν οι ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βελτίωση και αλλαγή ε, της λειτουργίας της Όλαφ. Τέλος, για να μπορέσει η Ένωση να συμβάλλει στην επίλυση των παγκοσμίων προβλημάτων, θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα κονδύλια και πώς ε, μεταφέρονται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική δράση. Κάνουμε και προόδου όμως, έχουμε και θετικά να πούμε. Τα κράτη-μέλη κάθε χρόνο κάνουν δηλώσεις για το πώς διαχειρίζονται ε, το προπολογισμό και αυτό είναι ένα παλιό πάγιο αίτημα των σοσιαλιστών. Και επίση για να μειωθούν τα σφάλματα, καλό είναι να ε, βελτιώνεται και να αυξάνεται η ανάκτηση των κονδυλίων. Παρ' όλα αυτά, ε, έχουμε κάποιες αμφιβολίες ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, απαλλαγή της. Σας ευχαριστώ. Περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρώτος και τώρα, ο δεύτερος αγωρητής, ο οποίος θα είναι η κυρία Γιάλα Σέντερ. Είναι η συγκήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενώπιόν μας έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ταμεία ε, περίοδος 7, 8 και 9 για την ε, χρήση του 2008 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η συγκυρία, διότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικέ μεταβολέ θεσμική ε, φύσεω, αλλά επίση έχουμε και όλε αυτέ τι διαφορετικέ κρίσει καταστροφές που έχουν γίνει στην παγκόσμια σκηνή και αυτό ε, δείχνει το πόσο είναι όλο ένα και πιο σημαντική η ευρωπαϊκή βοήθεια όσον αφορά το συντονισμό θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και ότι χρειάζεται να υπάρχει και διαφάνεια και έτσι όλοι οι πολίτες να συνεχίζουν να υποστηρίζουν ε, αυτή την, την, την πρωτοβουλία και να έχουν θετική άποψη για αυτήν. Βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα που είμαστε στην αρχή της περίοδου ισχύω της συνδίκης της Λισαβόνας ε, έχουμε την ε, υπηρεσία την, της εξωτερικής πολιτικής, επίσης έχουμε και την ε, ΚΕΠΑ, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι πιο καλή αυτή η εξωτερική βοήθεια, πώς θα είναι πιο αποτελεσματική, αλλά υπάρχουν και κάποια πάρα πολύ σημαντικά ερωτηματικά, γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτή η αποτελεσματικότητα που θέλουμε, αφού που να πετύχουμε με Κομισιόν και Ελληνικό Συνέδριο για την Αναπτυξιακή Ευρωπαϊκή Βοήθεια, είναι δυνατόν, λέγω, αυτή να δυναμητιστεί από το, το πόσο διφορούμε είναι οι αποφάσεις, ε, η, η διαχείριση να ε, είναι εμβαλωματική. Οπότε θα πρέπει η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους εκτροπές και το συντομότερο δυνατόν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με το πώς θα ισχύσει αυτό το καινούργιο σύστημα την αναπτυξιακή βοήθεια. Πρώτα-πρώτα τώρα, όσον αφορά αυτό το έργο που έχουμε ενωπιών μας, θα πρέπει να σας πω ότι χρειάζεται ε, να επαναλάβουμε ή θα πρέπει να εντάξουμε το αναπτυξιακό τομείο ε, σε αυτή την προσπάθεια για ε, έλεγχο και διαφάνεια. Οπότε και δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε ότι Κομισιόν και Κοινοβούλιο για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει αυτό το πάγιο έτοιμά μα να συνεχίσει να διατυπώνεται, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο την κοινή, τον κοινό προγραμματισμό, να έχουμε συντονισμό στη δουλειά μας και έτσι να μπορέσουμε ε, το δέκατο ταμείο να το περιορίσουμε σε συγκεκριμένους κλάδους και τομείς για να μην έχουμε επικαλύψεις, μην έχουμε ε, κάποιο είδους ε, υπονόμευση της αποτελεσματικότητας των μη κυβερνητικών οργανισμών που δουλεύουν επί τόπου. Δηλαδή είναι δύσκολο αυτό, είναι το εργαμό του κύκλου. Αλλά ελπίζουμε ότι σε συνεργασία με την Κομισιόν θα τα καταφέρουμε επίση. Θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα, μια που ήταν θετική η δήλωση αξιοπιστία εκτό από εκεί που έχουμε ε, κάποια έξοδα τη ε, Κομισιόν. Δεν είναι βέβαια πολύ μεγάλα τα σφάλματα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ε, επιφέρουμε κάποιες ε, βελτιώσεις όσον αφορά τις, ε, το, το, μέγεθος του σφάλματος και για τις πληρωμές και για τις υποχρεώσεις. Και για άλλη μία φορά δεν μπορεί το συνέδριο να έχει προσβασιμότητα σε κάποιο είδους τεκμηρίωση όσον αφορά κάποιους διεθνείς φορείς. Άρα θα πρέπει να υπάρχει κάποια αποκρυσταλλωμένη μέθοδος για να υπάρχει προσβασιμότητα σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις και να μην έχουμε προβλήματα έλλειψης διαφάνειας. Επομένως, το κλείσιμο του Ευρωδομού Ταμείου ε, ε, ήταν ε, τα πράγματα χωρίς πρόβλημα, έγιναν οι μεταφορές στο ένατο και μόνος θα πρέπει από τον Ιούλιο του 2008 να δούμε το ότι καλά τα πήγε το 10ο Ταμείο και επίσης το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την ρευστοποίηση των πληρωμών που εκκρεμούσαν. Επίσης προβληματιζόμαστε όσον αφορά διακόπτει ο Πρόεδρος αυτά τα οποία δεν καλύπτονται από την δήλωση αξιοπιστίας λέει η, ε, η και ότι θα πρέπει τελικά αυτό να καλυφθούν από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Μπάρτ Στάση έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αναρωτήθηκα τι εστί απαλλαγή. Η απαλλαγή είναι μια διακασία και κοινοβουλευτική και δημόσια. Μια δημόσια ε, κριτική εξέταση των δημοσίων οικονομικών και τη διαχείριση. Και αυτό έκανα για το Κοινοβούλιο για το 2008. Και ως μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά και οι πολίτες πλέον έχουν καλύτερη αίσθηση, καλύτερη αντίληψη για την ιδιαίτερη οργάνωση, την αναθιάρθρωση, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, οι πολίτε έχουν το δικαίωμα να ξέρουν τι γίνεται με το προπολογισμό μας, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Το 2008 1,4 δις ήταν ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Για το 2011 μάλλον 1,7 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Είναι ε, σημαντική η διαδικασία και σημαντική η δουλειά της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ε, γιατί αν έχει ένα κριτικό βλέμμα ε, οδηγεί σε προόδους στο παρελθόν το είδαμε αυτό. Ε, προέκυψε το καθεστώς των βουλευτών και το καθεστώς των βοηθών, ακριβώς επειδή το ζήτησε η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Επίσης, με κριτικό ε, βλέμμα είδαμε τι γίνεται με τα κτίρια στο Στρασβούργο. Οδηγήσαμε στη δημιουργία της διαδικασίας ΙΜΑΣ ε, για την οικολογική μας ε, στάση. Όλα αυτά είναι θετικά νέα, είναι καλά νέα. Μέσα σε μία τριετία ακριβώς μειώσαμε κατά 25% το, την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. 100% πράσινο ρεύμα έχουμε τώρα. 17% ε, μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Ε. Επίσης, 50% ε, μείωση των αποβλήτων με ανακύκλωση. Και στην έκθεση έχω βάλει και την έννοια των λεγόμενων κινδύνων υπόλοιψη για τη φήμη του Κοινοβουλίου. Γιατί ε, μπορεί με λίγα χρήματα, ε, αν χρησιμοποιούνται λάθος, να ε, υποστεί σοβαρή ζημία η φήμη και η υπόλοιψη του Κοινοβουλίου και το κύρος του. Επίσης, έχουμε διαχείριση κινδύνου. Ε, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με το έργο αυτό και το προσκαλώ να έρθει στις διάφορες επιτροπές για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο ε, ατασταλιών και ε, κακής χρήσης των χρημάτων στο Κοινοβούλιο. Μεγαλύτερη διαφάνεια λοιπόν, γι' αυτό ζητώ ένα σύστημα με ελέγχους και εξισορρόπηση, περισσότερη ευθύνη και αίσθημα ευθύνης. Προτείνω λοιπόν κύριε Πρόεδρε να σας δώσουμε την απαλλαγή. Δεν είδα μεγάλα σκάνδαλα, μεγάλες απάτες, μεγάλες ατασταλίες. Παραμένει όμως κριτική η έκθεσή μου και θέλω να δείξω ότι μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Η έκθεσή μου έχει στόχο να φροντίσει αν το 2014 όταν πάμε ξανά στις εκλογές να μην έχουμε σκάνδαλα ούτε μεγάλα ούτε μικρότερα και να μπορεί, να μην μπορεί κανείς να μας προσάψει τίποτα και να μην έχουμε κακά σχόλια στον τύπο και περίεργα δημοσιεύματα. Στην έκθεσή μου ε, ασχολήθηκα με το Γενικό Γραμματέα και ε, με τη διοίκηση για να τους βοηθήσω. Επίσης ε, αναφέρθηκα σε ορισμένα σημεία που χωλένουν. Ο Γενικός Γραμματέας ε, κάνει δηλώσεις κάθε χρόνο ε, με βάση τα όσα του λέγουν οι γενικοί διευθυντές. Εγώ θέλω και μια τρίτη γνώμη. Το σύστημα των δημοσίων προμηθειών, ας πούμε, είναι ένα θέμα που ενέχει πολλούς κινδύνους και θα πρέπει να το ξαναδούμε. Επίσης, διαπιστώνω ότι 121 εκατομμύρια αναλογιστικό έλλειμμα έχει το Ταμείο, το Επικουρικό Συνταξιοδότηση των Βουλευτών. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό σε σχέση με τα χρήματα των φορολογουμένων. Ε, προσπάθησα να συνεργαστώ καλά με του σκιώδει ηγητέ μου. Πολύ επικοδομητικέ οι τροπολογίε του. Λυπάμαι που κάποια στιγμή το Λαϊκό Κόμμα ζήτησε με 50 τροπολογίες να ε, ε, ε, διαγραφούν ορισμένες παράγραφοι ε, της έκθεσής μου κατόπιν ε, πίεσης που άσκησαν κύκλοι της διοίκησης. Λυπάμαι γι' αυτό. Εγώ θέλω να είμαι θετικός και επικοδομητικός σε αυτή την έκθεση και αυτό προσπάθησα να κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, γενικώ θα μπορούσε να πει κανεί ότι για όλα τα θεσμικά όργανα τα οποία καλύπτονται από την έκθεσή μου, ελεγκτικό συνέδριο, δικαστήριο, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, Διαμεσολαβητής, επόπτη τη προστασία των δεδομένων σε όλα αυτά τα θεσμικά όργανα, λέω, διαπιστώθηκαν καλύτερε επιδόσει. Βέβαια η κατάσταση απέχει από να χαρακτηριστεί τέλεια. Ε, το Συμβούλιο βέβαια προσφύγει τα πιο πολλά προβλήματα. Εδώ η κατάσταση δέχεται πολλές βελτιώσεις όσον αφορά τον προπολογισμό. Και αποφάσισα να αναβάλω την απόφαση χορήγησης της απαλλαγής για το Συμβούλιο. Αυτή η πρότασή μου υπευλήθη στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών και έγινε αποδεκτή. Πέρσι, οι συντονιστές της Επιτροπής είχαν συναντηθεί με την Προεδρία και είπαν ότι θεωρούνται πάρα πολύ θετικά τα βήματα βελτίωσης τη κατάστασης, όμως ακόμα εκκρεμούν κάποια προβλήματα. Αυτά πέρσι ε, όσον αφορά το Συμβούλιο ε, και στα ερωτήματα που έθεσαν δεν έδωσαν ικανοποιητικές απαντήσεις. Και γι' αυτό οι συντονιστέ από όλε τι πολιτικέ πτέρυγες του Κοινοβουλίου συμφώνησαν μαζί μου όταν αποφάσισα να αναβάλω την απόφαση χορήγησης τη απαλλαγή. Υπάρχουν κάποια θέματα της και ΠΑ, τα οποία ακόμα πρέπει να ξεκαθαριστούν, κάποια θέματα εκτός προπολογισμού, κάποια άλλοι λογαριασμοί, εντάλματα πληρωμής. Να δούμε πώς θα γίνει η καθάριση αυτών των εργασμών που εκκρεμούν. Επίση, έχουμε και κάποιε απαντήσει του Κοινοβουλίου που δόθηκαν όχι επί τη βάση τη τρέχουσα χρήση, αλλά τη προηγούμενη. Και το Λιγδό Συνέδριο επέσυρε την ε, προσοχή μα σε κάποιε αντικανονικότητε όσον αφορά του προκυρηθέντε διαγωνισμού. Γι' αυτό και αποφανθήκαμε ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να βελτιώσει τι συμπτώσει αυτέ τη ε, υποθέσει. Έχουμε σε πολλά θέματα που έχουν μαζευτεί και από μένα ξεκαθαριστούν. Έχουμε μια ειδική υπηρεσία με, με, ελέγχει που αφορά τους ελέγχους να δούμε αν η κατάσταση θα βελτιωθεί. Να δούμε αν οι επιδόσεις ήταν καλύτερες από πέρσι δηλαδή. Πάντως ακόμα έχει πάρα πολλές επιφυλάξεις στο ελληνικό συνέδριο όσον αφορά ε, την, την υποβολή των ε, δηλώσεων του οικονομικού συμφέροντος. Μάλλον έχει γίνει ορθή διαχείριση των οικονομικών του Ελληνικού Συνεδρίου, αλλά ακόμα υπάρχουν κάποια θέματα, ακόμα θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, ίσως θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μελών του Ελληνικού Συνεδρίου. Τώρα να σας πω για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έγινε έλεγχος από το Ελληνικό Συνέδριο. Οι λογαριασμοί ήταν εντάξει, όμως και εδώ η κατάσταση επιδέχεται βελτίωση. Θα πρέπει όλοι οι δημοσιομικονισμοί να εφαρμόζονται το ίδιο για όλα τα θεσμικά όργανα. Ευτυχώ υπάρχει βέβαια και αυτή η διοικητική συνεργασία. Υπάρχει συνεργασία διοικητική μεταξύ ΟΚΕ και Επιτροπής Περιφερειών. Υπάρχει εναρμόνιση σε κάποια θέματα που έπρεπε να γίνει και αυτό είναι θετικό. Και υπάρχουν κάποια προβλήματα μεταξύ διαμεσολαβητή και Επιτροπής Περιφερειών. Με κατακλείδη τα προβλήματά μα περιορίζονται στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να σεβαστούμε το χρονικό όριο του χρονικού περιορισμού, λέει και σα ευχαριστώ πάντω για όσα μα είπατε για την έκθεσή σα. Και από ό,τι μου λένε, ε, ήρθαν οι συνεργάτε μα σε επαφή με του επικεφαλεί των ιδιωτικών γραφείων του Πρόεδρου του Ελληνικού Συνεδρίου και σε σχέση με τις συζητήσεις που έγιναν το 2008 και 2009 ε, διαπιστώθηκε ότι ούτε τότε είχαν έρθει εκπρόσωποι του Ελληνικού Συνεδρίου αλλά ούτε τότε είχαν έρθει και εκπρόσωποι του Συμβουλίου ούτε από τον όργανο ούτε από το άλλο είχαν παραστεί τότε εκπρόσωποι κατά τη σχετική συζήτηση Ο κύριος Καλτέρα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, έχει τονίσει ότι η θέση του Ελληνικού Συνεδρίου είναι ότι για τεχνικά θέματα παρήσατε συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελληνικού Προπολογισμού. Αλλά δεν συμμετέχει στις πολιτικές συζητήσεις στην Ολομέλεια. Και είπε ο πρόεδρος Καλτέρα ότι προτίθεται να τις επαφή μαζί μου σήμερα και θα εξηγήσει τη θέση που αφορά το ελεγκτικό συνέδριο για τα θέματα της απαλλαγής. Επομένως, αυτό κοιτάξαμε να δούμε τι έγινε κατά τις τελευταίες συζητήσεις, τις τελευταίες δύο χρονιές. Δεν ήταν εδώ. Αυτό για ενημερωσή σας. Ίσως θα πρέπει να φροντίσουμε να το οργανώσουμε αλλιώς του χρόνου. Και ίσως θα πρέπει να έρθουν. Φυσικά και έχουν ενημερωθεί για την σημερινή συζήτηση. Αλλά ούτε πέρυσι το πρόβλημα είχαν παραστεί. Οκτώβριο και Νοέμβριο πάντως, οπωσδήποτε θα είναι εδώ, διότι τότε και θα εισηγηθούν τα θέματά τους, την εκθεσή τους. Να, μάλιστα, έχετε διαδικαστικό. Το έλαβα υπόψη. Ο κύριος Γκέρμπραντι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να δεχτώ πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο απουσιάζει, αλλά αυτό που μας είπατε τώρα για την απουσία του Συμβουλίου και τα προηγούμενα έτη ε, υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό και όχι συγκυριακό. Χαρακτηρίζει αυτό τη συμπεριφορά του Συμβουλίου απέναντι στην υπεύθυνη ε, διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και αυτό ξύνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Για το λόγο αυτό λοιπόν, για να στείλουμε ένα σαφέστατο μήνυμα από το Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο, θα πρότεινα το κεφάλαιο της απαλλαγής του Συμβουλίου να αναβληθεί και η συζήτηση και να μην συζητήσουμε καθόλου την απαλλαγή για το Συμβούλιο. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Τσανέρσκι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δώσατε όλες αυτές τις πληροφορίες σχετικά με την αποσία του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι τώρα βρούμε, ε, ενεργούμε με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας και ο ρόλος μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βελτιωθεί και επεκταθεί. Οπότε, από πολιτική άποψης, θα έπρεπε να αναμένουμε τους εκπροσώπους του Συμβουλίου εδώ. Όπως είπε και ο συνάδελφο πριν από μένα, πρόκειται για συζήτηση μεγάλη σημασία για τους φορολογούμενους μας, για τους ψηφοφόρου μας. Νομίζω πως εάν το Συμβούλιο Συγγνώμη, νομίζω πως το Συμβούλιο κάνει λάθος που αγνοεί και παραμελεί αυτή τη συζήτηση γιατί συμφωνώ ότι θα πρέπει να καθυστερήσουμε τη συζήτηση της απαλλαγής για το Συμβούλιο και να ναι. τονίσω ακόμα μια φορά ότι το Συμβούλιο δεν ε, ενεργεί, ενεργήσε επικοδομητικά στη συνεργασία μας όταν συναντηθήκαμε με τους συντονιστές στην Επιτροπή Προπολογισμού και πιστεύω πως η αποσία του σήμερα αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι δεν έχουν καθόλου επικοδομητικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ παίρνω τη θέση σας, η κυρία Χέρτζοκ τώρα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ε, γίνεται η διαδικασία απαλλαγή και ψηφίζουμε από αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει πλήρω την ευθύνη για το 2008. Οπότε είναι η στιγμή όπου εμεί αναλαμβάνουμε την ευθύνη και για όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, για το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τους διάφορους οργανισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία. Ωστόσο, εγώ συμφωνώ να συνεχίσουμε με τη συζήτηση και μην, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια αντικειμενική, ένα αντικειμενικό λόγο. Δεν είναι τόσο εύκολο να έρθει κανεί εδώ από το Ιν Ισπανία. Το ξέρω γιατί και εγώ ήρθα από το μέσο Μπακού και Μαδρίτη σε μέσο τρένου, με τρένο μάλλον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταξιδέψει κανεί και Εν πάση περιπτώσει, το Μάιο φαντάζομαι πως θα δείξουν το ενδιαφέρον τους ε, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας όλα τα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ, συνάδελφος Οντί. Oui, ναι, Πρόεδρε, έχουμε τη συνήθεια να βλέπουμε άδεια τα έδρανα του Συμβουλίου. Δεν είναι η πρώτη φορά, ας μην είμαστε ε, υποκριτές. Ε, εκφράζω το λύπημα λοιπόν ακόμα μια φορά. Εγώ είμαι υπέρ του να συνεχιστεί η συζήτηση. Πιστεύω εξάλλου ότι με την επιφύλαξη της γνώμης της δικής σας γραμματείας δεν έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη. Την γκρίναμε όταν ξεκίνησε η Ολομέλεια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επαναλάβουμε την λύπη μας για την απουσία του Συμβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, Λοιπόν, Συμβούλιο και Ελεγκτικό Συνέδριο σήμερα αποσιάζουν. Σαφώς ε, και θα δηλώσουμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας για το μέλλον προς τα δυο αυτά σώματα. Θα τους πω ότι θα θέλαμε να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια τέτοιων συνεδριάσεων. Επίσης ε, θα μιλήσω προσωπικά στον Πρωθυπουργό Σαπατέρο που προεδρεύει αυτή τη στιγμή και Α, θαύμα έγινε. Θαύμα, μόλις ήρθατε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Βλέπετε, συνάδελφοι. Συνάδελφοι, ε, μόλις λέγαμε ότι πόσο δυνατοί είμαστε μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, φανταστικό. Μέσα σε λίγα λεπτά εμφανίστηκε το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. προεδρεύοντα το Συμβουλίου. Και βέβαια θα έρθω σε επαφή με τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου. Γιατί σίγουρα είναι απαραίτητο να είναι παρόντας κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Σήμερα θα τους πάρω όλους τηλέφωνο. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ να κρατάτε το χρόνο σας, το χρόνο ομιλία σας. Η κυρία Βερονίκ Ματιέ, η συγγήτριά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, χαίρετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλώ ενώπιόν σας. Καλημέρα σας. Από το 2000 μέχρι το 2010 διαπιστώνουμε αύξηση κατά 70% των κοινοτικών ε, εισφορών στις ε, περιφερειακές υπηρεσίες ε, το 2000 ήταν εργαζόμενοι 1.219 στις υπηρεσίες αυτές και σήμερα 4.794 ε, χωρίς να μιλούμε για την υπηρεσία ανασυγκρότηση που έκλεισε το 2008 και θα ψηφίσουμε την τελευταία απαλλαγή τη στις Βρυξέλλες. Αυτή η γενική πρόοδος μπορεί να είναι εντυπωσιακή, ωστόσο κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου 2000-2010 είχε να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις η Ένωση. Δύο διευρύνσει καταρχήν το 2004-2007, 12 νέα κράτη-μέλη και άλλε προκλήσει. Ε, ε, απασχόληση, εναέρε ασφάλεια, ασφάλεια γενικότερα, μετανάστευση ε, και κατάρτιση. Και δημιουργήθηκαν αυτοί οι οργανισμοί για να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες. Με την πραγματογνωμοσύνη τους συνεισφέρουν στην πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτές τις τεράστιες προκλήσεις. Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται στενά για τα θέματα αυτά και οι οργανισμοί αυτοί είναι ε, κατεξοχήν ε, χώροι ανταλλαγής απόψεων. Και επειδή είναι αποκεντρωμένοι οι οργανισμοί αυτοί, ε, έρχεται η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες και αποκεντρώνει και τη δράση της. Έχει αυξηθεί λοιπόν και ο αριθμός των οργανισμών και των υπηρεσιών αυτών και ο προϋπολογισμός και τους φέρνει ενώπιον των ευθυνών τους και ω προ ε, τη δημοσιονομική διαχείριση και το Κοινοβούλιο έχουν αντίστοιχε υπηρεσίε και το Ελεκτικό Συνέδριο και ο Ιστορικό Έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζονται όλοι αυτοί η ενίσχυση για να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα ε, τι υπηρεσίε αυτέ, χωρί αυτό να σημαίνει ότι οι ίδιε δεν έχουν ε, ευθύνη. Σε ό,τι αφορά την απαλλαγή του 2008, θα ήθελα να θυμίσω τα πάγια προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι δημόσιες προμήθειες και ανάθεσή τους, η ε, μη ρεαλιστική διαδικασία επιλογής και μη διαφανής διαδικασία επιλογής του προσωπικού, ε, ακύρωση πιστώσεων, μη απορρόφηση πιστώσεων και ε, έλλειψη συγκεκριμένων στόχων. Επίσης διαπιστώνουμε ότι παρά τις προσπάθειες που ε, καταβάλουν οι οργανισμοί αυτοί δύσκολα μπορούν να εφαρμόσουν το δημοσιονομικό κανονισμό για κάποιους οργανισμούς μιλώ που είναι μικροί, οι πιο μικροί οργανισμοί δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις βαριές διαδικασίες που τους επιβάλλει ο κοινοτικός κανονισμός. Ε, θα ήθελα εδώ να σας ε, παραπέμψω στις ε, αποφάσεις τα συμπεράσματα μάλλον της αντίστοιχη ομάδας εργασίας. Ε, ωστόσο, οι δυσκολίες αυτές δεν ε, θέτουν ένα αμφιβόλο τη συμφωνία για την απαλλαγή του 2008 για το, ε, ε, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία τα πράγματα διαφέρουν. Μπορεί να έχουν γίνει εκεί ε, βελτιώσεις σε σχέση με το 2007 στη ΣΕΠΟΛ. Οι εσωτερικοί όμως οικονομικοί έλεγχοι που έχουν ε, γίνει έχουν βρει κατάφορες ατασταλίες στην οικονομική διαχείριση γι' αυτό ζητούμε αναβολή της απαλλαγής. Τελειώνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω τις που κάνουν κάποιε κοινοτικέ υπηρεσίε για τη βελτίωση τη λειτουργία του. Ορισμένε, αυθόρμητα προχώρησαν ε, σε κανόνε που ε, αξίζει να του υπογραμμίσουμε και να του καθορίσουμε. Η ΕΦΣΑ, για παράδειγμα, για τη διατροφική ασφάλεια που είναι πάρα πολύ ε, ε, καλή ε, στη διαχείριση κινδύνου και στο συντονισμό. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος επίσης έχει κάνει ένα σύστημα ελέγχου για το πώς χρησιμοποιούνται σε πραγματικό χρόνο τα κονδύλια τους και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση, τελειώνω πρόεδρε, της εργασίας έχει ένα δικό του σύστημα παρακολούθησης. Βεβαίως καλώ τις υπηρεσίες να ακολουθήσουν αυτή την ατραπόκηση. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για την έκθεση και την εισήγησή σας, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα απευθυνθούμε εις τον Επίτροπο. Ουλάς... Κύριε Σεμέτα, έχετε το λόγο. Thank you, President. Mr. President, Secretary of State, uh, Rapporteurs, Honorable Members. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα πρέπει να ευχαριστήσω την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και συγκεκριμένα τον εισηγητή, τον κύριο Λιμπεράτσκι, αλλά και τους άλλους συνεισηγητές για τις σχετικέ εκθέσεις. Τη ευχαριστώ επίσης και για την απόφασή σας να χορηγήσετε την απαλλαγή για τη χρήση του 2008. Επίσης, ευχαριστώ και την κυρία Γιάλα Σέντερ για τη δική της έκθεση όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού του Ταμείου Ανάπτυξη, αλλά και την κυρία Ματιέ για αυτή την τόσο παικτική ανάλυση όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ. Τώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία χορηγή της απαλλαγής. Ήταν ε, εντατική και έντονη η εργασία μας, αλλά ήταν και επικοδομητικός ο διάλογος μεταξύ θεσμικών οργάνων. Ο στόχος της Επιτροπής είναι να έχουμε μια δήλωση από το Ελληνικό Συνέδριο που να είναι απερίφραστη και χωρίς ε, προϋποθέσεις και επιφυλάξεις. Ήδη έχουμε σημειώσει πρόοδο. Έχουμε επιφέρει κάποιες ε, απλουστεύσει, καλύτερη διαχείριση, καλύτερο έλεγχο ε, για την περιοδο του 2017 2007-2013. Επίσης και κάποια προγράμματα δράσης και έτσι φάνηκε πόσο θετικές επιπτώσεις υπάρχουν από τη δουλειά μας και θα μπορέσουμε να επιφέρουμε σημαντικές αλλαγές με τα προγράμματα της νέας γενιάς για την επόμενη ε, περίοδο. Είναι κάτι το οποίο τώρα το εξεργαζόμαστε και έτσι θα έχουμε καλύτερα κριτήρια επιλεξιμότητας, έλεγχο των δαπανών και δαπάνες που να χαρακτηρίζονται από καλή ποιότητα. Πάντως, πάρα πολύ σύντομα, θέλουμε να έχουμε κάποια μετρήσιμη πρόοδο όσον αφορά την διαχείριση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και να περιορίσουμε τα θέματα ευθύνη, υπευθυνότητας και λογοδοσίας των εμπλεκομένων. Οπότε ο δικό ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πάντως γνωρίζουμε όλοι ότι δεν αρκεί το να επιταχύνουμε τον ρυθμό βελτίωσης των επιδόσεων. Θέλουμε καλύτερη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Θέλουμε ενεργά να βοηθήσουν και τα κρατη και το Ελληνικό Συνέδριο. Δεν θα περιμένουμε να τροποποιηθεί ο γεμεσονικός κανονισμός. Καλούμε από τώρα τα κρατη να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ακριβώς όπως ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Και από τώρα να ληφθούν κάποια μέτρα για να βελτιώσουμε την ε, διαχείριση των πόρων. Βεβαίω, το Ελληνικό Συνέδριο έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά και αυτό τονίστηκε και στην δήλωση αξιοπιστίας που αφορά τα της Κομισιόν, τη διαχείριση των χρημάτων. Σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς μας. Και δεν μπορούμε να παραθέσουμε κάτι πάρα πολύ θετικό. Το ότι στο άμεσο μέλλον το Ελληνικό συνέδριο θα κάνει διάκριση μεταξύ των τομέων ανάλογα της διαφοράς κινδύνου σφάλματος. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχα διαφορετικά συστήματα ελέγχου. Και όλα αυτά θα υλοποιηθούν και θα ισχύσουν και κατά την περίοδο 2007-2013. Και εσείς συμφωνήσατε και έχουμε και αυτή τη νέα έννοια του ανεκτού κινδύνου σφάλματος. Εμείς θα εκπονήσουμε και θα σας υποβάλουμε μια, ένα, κατάλογο με θέματα εργασιών για την περίοδο 2010 και μετά. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα μειωθεί κίνδυνο σφάλματος και να πάμε στο 20% του προπολογισμού για το 2014 όσον αφορά αυτό που έχει ζητήσει το Ελληνικό Συνέδριο. Έγινε κοινό μα στόχο η βελτίωση τη οικονομική διαχείριση και η προστασία των εγγονών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, για αυτό το νέο πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα σας υποβάλουμε, αυτό το ζήτημα θα είναι στο επίκεντρο. Και όσα διατυπώνετε στο ψήφισμά σας θα τα λάβουμε υπόψη και περιμένουμε πώ και πώ την επιδομική συνεργασία μαζί σα. Σας ευχαριστώ. που μας παρουσιάσατε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το οικονομικό έτος 2008 στους τομείς πολιτικής ε, που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Εξωτερικών οι πληρωμές έφτασαν περίπου τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. διαπιστώνουμε ότι η κατηγορία 4 υποχρηματοδοτείται ήδη από το παρελθόν. Διαπιστώνουμε κάποιες ε, ε, μικρές ε, ε και το ελεκτικό συνέδριο ε, τα ελέγχει αυτά αποσπασματικά, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τα προγράμματα είναι πολυετή τα περισσότερα και το ελεκτικό συνέδριο τα εξτάζει ετησίως αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν ε, κάνει λόγο το ελεκτικό ε, συνέδριο ούτε για απιστία ούτε για απάτη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εγκαίρως να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης και να ε, λογοδοτεί. Γιατί είναι λυπηρό να είναι ανεπιτυχή τα προγράμματα ή να μην καταβάλλονται οι πόροι εγκαίρως. Αυτό διακυβεύει την επιτυχία της εξωτερικής μας πολιτικής. Καλή λοιπόν η συνεργασία μας και παρελθόν και καλή ε, της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Από ό,τι φαίνεται αρχίζουν να αποδίδουν τα μέτρα που ελήφθησαν για την αλλαγή. Η ε, έκτακτη έκθεση ε, πρόοδου για την ε, Τουρκία κάνει λόγο για βελτίωση με το νέο προενταξιακό μέσο από το 2007 και μετά. Επιπλέον, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για τη χρήση που κάνουν οι δικαιούχοι των κοινωτικών κονδυλίων με ευεξία να προσαρμόζουμε κάθε φορά την κατάσταση για να επιτυχάνουμε τους στόχους μας. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει το δημοσιονομικό κανονισμό ε, την ίδρυση τώρα ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Από πλευρά όμως ΑΦΕΤ μπορώ να συστήσω την απαλλαγή για το έτος 2008 σε γενικές γραμμές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Η κυρία Γκρέσλε έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύον, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ενδιαφέρον το πρωινό σήμερα. Κανονικά θα ήθελα να πω κάτι άλλο τελείως. Δεν θα το κάνω. Δεν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε έτσι αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ για να το ξεπεράσουμε. Ποιο είναι το γεγονός. Η απαλλαγή αυτή δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ε, απαλλαγή ούτε από το Κοινοβούλιο ούτε από τα άλλα θεσμικά όργανα. Η μόνη που παίρνει σοβαρά υπόψη της τα θέματα αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την αφορά άλλωστε το θέμα πάρα πολύ. Ε, για τα άλλα θεσμικά όργανα το θέμα της απαλλαγής δεν ε, ρορίζεται από τις συνθήκες. Και τι θα γίνει με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης αν γίνει θεσμικό όργανο και αυτή θα απουσιάζει στο μέλλον ούτε καν το θεωρούν σκόπιμο και χρήσιμο και αναγκαίο να παρευρίσκονται για να ακούν τι έχει να του πει το Κοινοβούλιο ως νομοθέτης ε, για τον προπολογισμό. Το ε, Συμβούλιο παρευρίσκεται, εξαίρεση λαμπρή αυτή, όπως και η Σουηδική Προεδρία πέρυσι. Είναι βασικό δικαίωμα του Κοινοβούλιου η απαλλαγή. Προσοχή, ε, προειδοποιώ να μην κάνουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης θεσμικό όργανο, γιατί εκεί θα τελειώσει και η επιρροή μας. Δεν θα έρχονται στις συζητήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου σήμερα το πρωί και για το γεγονό ότι έρχεται σε επαφή με του ομολόγου του. Τι να το κάνουμε να έχουμε δικαίωμα απαλλαγή, αν δεν μα παίρνουν στα σοβαρά και αν δεν είναι αγκασμένοι, υποχρεωμένοι άλλοι να παρευρίσκονται να ακούνε αυτά που έχουν να του πούμε. Θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό το θέμα της απαλλαγής και δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση όσο έχει. Επευκαιρία να απευθυνθώ και στο Συμβούλιο. Μετά τη Λισαβόνα το Συμβούλιο έγινε θεσμικό όργανο και η Προεδρία του Συμβουλίου. Θα πρέπει ε, επιγόντως αυτό να μεταφραστεί και στο δημοσιονομικό δίκαιο. Θα πρέπει να είστε ε, αρμόδιοι για τα οικονομικά τα δικά σας και για το Συμβούλιο και για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Παρακαλώ να νομιμοποιηθεί, να τακτοποιηθεί αυτή η κατάσταση επιγόντως. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρος, κυρία Γκρέσλε. Η κυρία Χάουκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα μόνο σημείο θα ήθελα να φέρω εγώ, ένα σημείο που είναι σκέτο σκάνδαλο. Το κέντρο λέει για την πρόληψη και έλεγχο νοσημάτων στη η ECDC. Από το Μάιο του 2005 άνθρωποι με πολύ υψηλά προσόντα ε, ε, δουλεύουν σε ένα απόλυτα εχθρικό περιβάλλον. Μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει η Σουηδική Κυβέρνηση να υπογράψει σύμβαση για την έδρα που ήθελαν οπωσδήποτε να την πάρουν. Όπω όλα κράτη-μέλη παλεύουν και αγωνίζονται για να έχουν οπωσδήποτε ένα οργανισμό, μια τέτοια υπηρεσία. Δεν έχουν ούτε καν ε, αριθμό ε, που χρησιμοποιείται ε, ε, από την κοινωνική ασφάλιση ο προσωπικός αριθμός του καθενός ε, ε, για να έχουν σχέσεις οι πολίτες με τις αρχές. Δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά του σχολείο, να πάνε σε νοσοκομεία, να βάλουν ρεύμα, νερό, τηλεόραση στο σπίτι τους εφόσον δεν έχουν αυτό τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης που έχει ο κάθε πολίτης που ζει στη Σουηδία και θα μπορούσα εδώ να πω πολλά ακόμα. Υπάρχουν πολλά δικαιώματα, βασικά δικαιώματα και θεμελιώδη, τα οποία αρνούνται ε, ορισμένοι στους εργαζόμενους ε, στη Στοκχόλμη. Και όλα αυτά κατέληξαν στην Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, είναι αφόρητη η κατάσταση. Ο πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Ο κύριος Φαντεκάμπ έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊ... της Επιτροπής μας ΙΜΚΟ για το 2008 δεν έχει και πολλά ακόμα να πούμε. Στην ε, Επιτροπή και στις εκθέσεις αυτά που είπαμε διευκρίνησαν πολύ την κατάσταση. Το 2008 είχαμε υπό απορρόφηση των πόρων στο Solvit αυτό όμως το 2009 και το 2010 θα διορθωθεί. Θα ήθελα να παρακαλέσω λοιπόν τον Επίτροπο να φροντίσει να γίνεται καλή χρήση του προϋπολογισμού για το Solvit. Εφόσον υπάρχει προϋπολογισμός υποθέτω ότι με ευθύνη ε, δαπανάτε αλλά δεν έχουμε πολλές πληροφορίες σχετικά. Και ίσως να πω και λίγα λόγια για την ε, οδηγία για την παροχή υπηρεσιών του Δεκεμβρίου 2009 και εδώ χρειάζεται ε, ενημέρωση και καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα άλλο θέμα αφορά τον ουσιαστικό τελωνιακό έλεγχο των κρατών μελών. Δεν είναι ένα θέμα που μας απασχολεί άμεσα τώρα, αλλά βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν ελέγχουν την εισαγωγή αγαθών όσο θα έπρεπε και θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το ξανασκεφτεί, να το συζητήσει με τα κράτη-μέλη να ελέγχουν σωστά την εισαγωγή επορευμάτων στην Ένωση. Τέλος, Πρόεδρε, κάτι που είπα πολλοί συνάδελφοι και ο ίδιος ο Επίτροπος, οι κανόνες του προπολογισμού σε πολλά σημεία είναι ακόμα πάρα πολύ περίπλοκοι και αυτό σημαίνει ότι και οι μηχανισμοί ελέγχου ε, είναι επίσης περίπλοκοι. Και ε, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε ε, προσπάθεια για απλούστευση και για βελτίωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιάλα Σέντερ, για ένα λεπτό παρακαλώ. το πρώτο κομμάτι το διαδικαστικό. έτσι θα το ζήταγα πριν. Θα ήθελα μέχρι τότε συζήτηση να μάθω εάν, όπως και το Συμβούλιο, πρόκειται να έρθει και αν, αν τους καλέσατε βέβαια εκπροσώπους του Ελληνικού Συνεδρίου Επίσης, θα πρέπει να δούμε εάν ε, είχε έρθει και το Συμβουλίο Σουηδική Προεδρία στη σχετική συζήτηση για την απαλλαγή. Από τώρα μπορεί να αρχίσετε να μετράτε το χρόνο όσον αφορά την απαλλαγή για τις μεταφορές. Πρώτα-πρώτα, πρέπει να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το πόσο έλαβε υπόψη η Κομισιόν αυτό το οποίο λέγαμε όσον αφορά τις πτώσεις πληρωμών και υποχρεώσεων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Σχεδόν πήγαμε στο 100%. Επίση, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι τα κράτη-μέλη να παράσχουν εγγύησει για επαρκή χρηματοδότηση από του εθνικού προπολογισμού. Επίση, θα πρέπει να επενθυμίσουμε και πάλι ότι πάντα υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη χρηματοδότηση για τα δίκτυα. Και επομένω θα πρέπει να δούμε για την περίοδο μέχρι το 2010 εάν ήταν επαρκή η χρηματοδότηση που έγινε. Πάντως, ο έλεγχος πήγε μια χαρά. Επίσης είναι πάρα πολύ θετικά τα αποτελέσματα όσον αφορά την νομιμότητα των, της διαχείρισης. Είχαμε βέβαια καθυστέρηση της προβλήψης του προσωπικού, αλλά είπε η Γενική ε, Διεύθυνση η Αρμόδη ότι πρόκειται να, να ενημερώσουν τη διαδικασία του σχετικά επίσης, πιστώσεις πληρωμών προς την ε, ασφάλεια των μεταφορών ήταν ε, κάτι το οποίο υστέρησε σε σχέση με τόσα ζήτησε το Κοινοβούλιο. Το ίδιο αφορά και τις πιστώσεις που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των ε, επιβατών. Γαλιλαίος και εκεί δεν είχαμε αρκετέ πληροφορίε ούτε και για τον τουρισμό. Ελπίζω ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα επιληθούν αυτέ οι αδυναμίε, αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιάλα. Τώρα έχει ζητήσει το λόγο ο κύριο Οντί. Διαδικαστικό έχετε. Διστάζω. Να παρέμβω ή όχι. Λυπούμε, αλλά θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω το Συμβούλιο και να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα, κύριε Υπουργέ, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήθιστε κύριε Πρόεδρε μετά την Κομισιόν να προτείνετε στο Συμβούλιο να πάρει το λόγο αλλά το Συμβούλιο ε, δηλαδή θα πρέπει να εκφραστεί πριν από την πολιτική συζήτηση. Ε, και ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να το ακούσουμε και να το ακούσουμε την αντίδρασή του στην θέση του εισηγητή που, είναι, που προτείνει την αναβολή της απαλλαγής για το Συμβούλιο. Θα συνεννοηθούμε με το Συμβούλιο αν θεωρεί σκόπιμο να παρέμβει. Ο κύριος Σούριαν για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η απαλλαγή είναι νομική πράξη από πλευρά Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Πρέπει να σα πω ότι δεν έχουμε καμία ένσταση όσον αφορά τη χορήγηση απαλλαγή. Όμω, εκτό από νομική πράξη, είναι και πολιτική πράξη. Και άρα θα πρέπει να δούμε αν καταφέραμε τόσο είχαμε τάξει ω στόχου για τη χρήση του 2008. Επίσης, να δούμε κατά πόσο πιάσαν τόπο τα όσα χρήματα δαπανίσαμε. Θα πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση τη πολιτική συνοχής. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ παρεξηγήσει για την πολιτική μας αυτή και σας επισημαίνω ότι τα λάθη πολλέ φορές προέρχονται από αμέλεια. Πολλές φορές το παρακάνουμε την ε, κριτική με τις επικρίσεις μας βεβαίως και το ελληνικό συνέδριο ε, διατυπώνει κάποιες επικρίσεις, με δουλειά του, αλλά θα πρέπει να πρέπει να πράγματα στις σωστές Δεν έχουμε ενιαίους δείκτες και ενιαία μεθοδολογία. Θα πρέπει να αποκτήσουμε. Αυτό αφορά και τους ρυθμούς απορρόφησης των πόρων. Αυτό πρέπει να το προσέχουν για την πολιτική συνοχή. Μόνο 32% των δαπανών προέρχονται από τα ταμεία. Όλα τα υπόλοιπα χρήματα ήταν χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν πριν έρθει το 2008. Να αποφασίσουμε επομένω και να καταλήξουμε στο τι έγινε το 2008 αν τα πήγαμε καλά ή όχι. πάντω, ε, όσον αφορά την απορροφητικότητα και απορρόφηση, μερικά κράτη δεν έφτασαν καν το 32%. Να δούμε τι έγινε, γιατί είχαμε τόσες καθυστερήσει, γιατί καθυστέρησε η Κομισιόν ή το Κοινοβούλιο. Προσπαθήσαμε από το 2008 και μετά να επιφέρουμε κάποιε απλωστεύσεις, να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Εμεί κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ε, τι κάνουμε στα κράτη-μέλη, τον είναι στο δικό του γήπεδο. Αυτοί να δούμε τι, τι κάνουν και τι θα κάνουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόριαντ. Ο κύριος Λόπης Αγγιλάρ τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ο κύριος Λόπης Αγγιλάρ απουσιάζει. κυρία Μπάουερ τότε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να θυμίσω ότι η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άρθρο 8 συγκεκριμένα προβλέπει την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και την προώθησή της. Αυτό είναι αρχή και θα πρέπει να τιμούμε τα όσα υπογράφουμε και συμφωνούμε σε όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και στη χορήγηση της απαλλαγής. Αυτή η αρχή θα πρέπει να βρίσκει εφαρμογή. Είναι απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να γίνει αυτό να έχουμε στατιστικά στοιχεία που ε, να ε, ε, περιγράφουν την κατάσταση. Διαπιστώνουμε με λύπη παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλουμε ότι δεν έχουμε τα στοιχεία που θα μας χρειάζονταν για να δράσουμε σε αυτή την κατεύθυνση για να ε, βρει εφαρμογή η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Αφορά αυτό δε διάφορους πολύ σημαντικούς ε, τομείς για την άρση των διακρίσεων, ε, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα που είναι ο εξής ίδρυση του Οργανισμού για την Ισότητα των Φύλων ε, διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις. Κανονικά το 2008 θα έπρεπε να αρχίσει να λειτουργεί ε, το κέντρο αυτό, ο οργανισμός αυτός και αρχίζει να λειτουργεί μόλις τον Ιούνιο του 2010. Αυτό ε, προκαλεί και τεράστια προβλήματα δημοσιονομικά. Δεδομένου ότι τα προγράμματα είναι πολυετή, ε, και το 2010 έχουμε την ενδιάμεση αξιολόγησή τους. Θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει ένα σύστημα που να επιτρέπει ε, ε, οι διάφορες θέσεις του προϋπολογισμού να εξετάζονται και με βάση την αρχή αυτή της ισότητας των φύλων. Και στον προϋπολογισμό λοιπόν να έχουμε αυτό το στοιχείο και να το εφαρμόζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Ο κύριος Μίτσελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από πλευρά τη πολιτική ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντική η απαλλαγή. Γιατί έτσι προστατεύουμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Ότι δηλαδή αυτά που πληρώνουν ε, πιάνουν τόπο. Έχουμε όσον αφορά το 0,7 του ΑΕΠ το οποίο ε, δίνεται ως συμβολή και θα πρέπει τελικά να ψυχιακή βοήθεια ε, να μην θέλουμε να είναι περισσότεροι ποσοτικά, αλλά να είναι καλύτεροι ποιοτικά και να δίνονται ευκαιρίες στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Οπότε, να δούμε τι θα γίνει στον την κυριότητα της γης, απλώς φυσικών προσώπων, κοινοτήτων και ολοκλήρων οικογενειών. Η φυματίωση, η ελωνοσία σκοτώνουν πάρα πολύ κόσμο στις χώρες. Και γι' αυτό και είπαμε τα τρία θεσμικά όργανα να δώσουμε το 20% από τους πόρους μας για υγεία και παιδεία. Πετύχαμε τους στόχους μας. Εγώ όποτε πήγα κάποια αποστολή στις αναπτυσσόμενες χώρες με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό το οποίο είδα. Εκεί οι νέοι μπορούν να καταφέρουν όσο καταφέρουν οι νέοι παντού. Άρα χρειάζονται ευκαιρίες και η παιδεία θα τους δώσει αυτές τις ευκαιρίες. Συμφωνήσαμε για αυτούς τους στόχους και τώρα θα πρέπει το σύστημα οικονομικού ελέγχου να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων αυτών, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να πω στο λίγο χρόνο ότι κατά τη γνώμη μου ο τρόπος, η λύση για το πρόβλημα αυτό της φτώχειας είναι το να κάνουμε κάποιες προσπάθειες για την ανακατανομή της κυριότητας της γης σε τις χώρες. Μιλάμε για ρυθμίσεις του 19ου αιώνα. Ε, αυτό ακόμα και στην Ιρλανδία είναι πρόβλημα. Αυτό σημαίνει δεξιακή βοήθεια. Να τους δώσουμε ευκαιρίες να επιτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ε, με τον κύριο Μίτσελ ολοκληρώνεται το κατάλογο των αγορητών εξ ονόματος των Επιτροπών και ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Ήτελε για τρία λεπτά. Παρακαλώ. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο που βρίσκεται σήμερα εδώ. Φυσικά Εκείνοι έχουν ευθύνη επίσης για τα χρήματα τα οποία εγκρίνουμε και γι' αυτό και είμαι πολύ ευχαριστημένος που είναι σήμερα παρόντες και που υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας. Για το Κοινοβούλιο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Στάς για την πολύ καλή συνεργασία. Η, βασικές, ε, η βασική ιδέα είναι ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι αρκετά ανοιχτό και διαφανές ώστε να μπορεί να αποκρούσει σκάνδαλα. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ε, την ε, χρήση των κονδυλίων, γιατί δεν είναι δικά μας χρήματα, δεν είναι δηλαδή του Κοινοβουλίου χρήματα, είναι τα χρήματα των φορολογουμένων και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε διαφανείς και να αναλαμβάνουμε τις ε, ευθύνες μας. Υπάρχουν ε, καλές αρχές στην έκθεση. Η ομάδα μου πιστεύει πως θα πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι, πιο συμπαγείς. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να μείνουν εκτός και ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στα πρακτικά ζητήματα. Ε, πάντως κάνουμε καλή δουλειά εδώ, να επιστιάσουμε στην, ε, στο νομοθετικό μας έργο που είναι η βασική μας εργασία εδώ. Έχουμε χώρο βέβαια για βελτίωση όσον αφορά την πολιτική περικτηρίων, να εντοπίσουμε τα προβλήματα στην έκθεση, γιατί αυτά είναι θέματα προσυζήτηση. Φαίνεται να, είμαστε, να έχουμε καθυστερήσει κάπως αυτή τη συζήτηση και χρειάζονται απαντήσεις οπωσδήποτε. Επιτέλους το Κοινοβούλιο κατάφερε να έχει ένα σαφές καθεστώς για τα μέλη του και για τους βοηθούς και αυτό είναι μόνο ένα βήμα στην πορεία. Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να αλλάξουν. Για παράδειγμα, τα προβλήματα πρόσβαση στο Στρασβούργο με το νέο καθεστώς εγώ πρέπει να επιστρέψω στο σπίτι μου κάθε φορά μετά το Στρασβούργο, αλλά είναι πιο εύκολο να πάω στις Βρυξέλλες. Είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση στην χώρα μου, στο Τούρτουλ της Φιλανδίας. Δεν έχω πια χρόνο, πρέπει να ξαναξεκινήσω και να ξανάρθω. Είναι δύσκολο λοιπόν να φέρει κανεί σε πλήρω τι ευθύνε του εδώ. Ε, δεν ξέρω, η Ρώμη, η Αθήνα είναι πιο εύκολα. Εγώ πολλέ φορέ προτιμώ να μείνω στι Βρυξέλλες και να αποφύγω όλη αυτή την ταλαιπωρία, καθώ και να, κάνω, να δουλέψω εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ήθελε. Ο κυρία Χέρτσο για τρία λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Στάς και να ευχαριστήσω και το ελεκτικό συνέδριο γιατί χάρη στην εργασία τους καταφέραμε να έχουμε μια συνολική εικόνα σε σχέση με το έργο του Κοινοβουλίου το έτος 2008. Είμαι επίσης ευγνώμων προς όλους τους συναδέλφους οι οποίοι με τις τροπολογίες τους έχουν βελτιώσει την έκθεσή μου. Σε ό,τι αφορά τα πραγματικά γεγονότα, Υπάρχει νομίζω μια ομοφωνία μεταξύ μας. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιήθηκε προπολογισμό το 2008 γιατί αφορά και του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε χρήματα από του φορολογούμενου και το ερώτημα είναι αν πράγματι χρησιμοποιήθηκαν τα ποσά αυτά βάσει των στόχων που είχαμε θεσπίσει εμεί ήδη. Έχουμε μια χρηματοοικονομική κρίση η οποία επηρεάζει όλου του πολίτε μα αυτή τη στιγμή Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το πώ θα δαπανίσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Οι προσδοκίε μα θα πρέπει να είναι ακόμα πιο υψηλέ έναντι ημών των ιδίων με ήττα παρά έναντι των άλλων. Αυτό είναι ένα θέμα αξιοπιστία για μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπενθυμίσουμε ότι η έλεγχή μα δεν είναι επαρκή αυτή καθεαυτή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπήρξε μια στα δαπάνηση των κονδυλίων και φυσικά σύμμορφη με τους κανόνες. Αυτό είναι δυνατό να γίνει μονάχα αν έχουμε ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχου το οποίο λειτουργεί με τρόπο ισχυρό. Εμείς θεωρούμε ότι ως σοσιαλιστές πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει λοιπόν, de facto, να ενισχύσουμε το σύστημα αυτό. Καλύτερη πρόληψη παρά η θεραπεία. Το ξέρουμε αυτό. Χρειαζόμαστε ένα στο εσωτερικό έλεγχο γιατί αυτό εξασφαλίζει και την ανεξαρτησία τη διοικητική διαχείριση. Με τον τρόπο αυτό θα βρισκόμαστε σε αρμονία με τι βέλτιστε πρακτικέ και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Φυσικά οι κανόνε αυτοί μόνοι του δεν μπορούν να εξασφαλίσουν του κατάλληλου εσωτερικού λογιστικού ελέγχου. Για το έτο 2009 χρειαζόμαστε, όπω ξέρουμε πολύ καλά, και περαιτέρω βελτιώσει για να έχουμε τέτοια συστήματα τα οποία είναι εύρωστα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τα συστατικά ενός τέτοιου συστήματος ελέγχου. Τίποτα το οποίο έχει φτιαχτεί από ανθρώπινα χέρια δεν μπορεί να είναι τέλειο. Πρέπει λοιπόν μετά από τον εσωτερικό έλεγχο να είμαστε προσεκτικοί και στη διαδικασία απαλλαγή. Θέλουμε να υποστηρίξουμε λοιπόν όλου του στόχου οι οποίοι θα θεσπίσουν εφικτού στόχου. Δεν θέλουμε όμω να έχουμε κάτι το οποίο θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και περαιτέρω νεφελώδει καταστάσει. Έχουμε προτάσει λοιπόν από τι πολιτικέ ομάδε. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου στον εσωτερικό του έλεγχο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο γιατί έχουμε τι δικέ μα ευθύνε. Ω ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, εμεί ακολουθούμε αυτέ τι οδηγίε ε, στην εργασία μα εάν και οι άλλες πολιτικές ομάδες θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας, παρακαλώ, είσαστε ελεύθεροι να το πράξετε. Γι' αυτό θέλω να δεχτείτε την έκθεση αυτή, να την υποστηρίξετε και να δώσετε την απαλλαγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Τσόγκο. Κύριος Γκερμπράντι για τέσσερα λεπτά. Καν... Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ είμαι μέγα υποστηρικτή ε, του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Genesis. Dance on the Volcano λέγεται ένα κομμάτι τους και το θυμήθηκα αυτή τη βδομάδα με την ηφαιστειακή τέφρα και τη σποδό. Όχι για να πάω στο ηφαίστειο να ε, χορέψω, αλλά μου ήρθε στο μυαλό ε, αυτό σήμερα το πρωί για την απαλλαγή του 2008. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, και πάλι δεν ξέρω αν θα πρέπει να το εγκρίνει. Και το εφέσιο αυτό δεν έχει ούτε λάβα, ούτε τέφρα, αλλά είναι γεμάτο δυσπιστία. Και είναι πολύ μεγάλη η πίεση στην Ευρώπη, πίεση επί του ευρώ, πίεση μεταξύ των κοινοτικών και των εθνικών ε, διοικήσεων. Αυτό που δεν μπορούμε εμείς όμως να ανεχτούμε είναι να εκραγεί το ηφαίστειο αυτό ε, λόγω κακής ε, δημοσιονομικής χρήσης, λόγω δυσπιστίας στα μάτια των πολιτών. Πώς γίνει αυτό να προληφθεί. Με ένα και μόνο τρόπο, διαφάνεια. Η βέλτιστη διαφάνεια παντού, σε όλα τα θεσμικά όργανα. Ε, για το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη και χαίρομαι που επιτέλους έφτασε το Συμβούλιο και παρευρίσκεται ακριβώς γιατί είναι η μεγαλύτερη πηγή ατασταλιών. Κάθε χρόνο διαπιστώνουμε ε, και νέε. Και καλό τα κράτη-μέλη επιτέλους ε, να λογοδοτούν κάθε χρόνο για τους κοινοτικού πόρους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ε, τα κράτη-μέλη ανθίστανται και εξακολουθούν να αντιδρούν. Τα δικά τους χρήματα με τον ίδιο τρόπο τα διαχειρίζονται. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο για τους πολίτες τους. Μεγαλύτερη διαφάνεια όμω χρειάζεται και για το κοινοβούλιο μας, για τι έχει δίκιο ο Μπαρτ και έχει κάνει μια πάρα πολύ κριτική έκθεση και ε, μιλάει για τις μεγάλες βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Ε, δεν ε, είναι τώρα η ώρα άρα για να ανοίξουμε τα παράθυρα διάπλατα και να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες και φορολογούμενους τι κάνουμε με τα χρήματά μας και πώς τα χειριζόμαστε υπεύθυνα, τα δικά τους χρήματα. Πριν από 40 χρόνια χρειάστηκε συμφωνία κυρίων για να ε, επικρατεί μια γενική ηρεμία. Τότε ήταν αυτό πάρα πολύ χρήσιμο για να μην υπάρχουν φασαρίες και ε, καυγάδες. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς θα πρέπει να λέμε ότι αυτά είναι πλέον απορχιωμένα και ε, δεν επικρατεί η ηρεμία ίσα ίσα στο μεταξύ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενηλικιωθεί ως θεσμικά όργανα και θα πρέπει ως ενήλικες να μπορούν ο ένας να ελέγχουν τον άλλον, χωρίς συμφωνία κυρίων. Και θα ήθελα να ρωτήσω το παρόν πλέον Συμβούλιο. Ε, πώς απαντάτε σε αυτό. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με καλό τρόπο να ελέγχει ο ένας τον άλλον χωρίς αυτή τη συμφωνία κυρίων. Πρόεδρε, χωρίς αυτή τη συμφωνία κυρίων και με αμοιβαία διαφάνεια μπορούν να χορεύουν ε, αρμονικά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, χωρίς να ε, φοβάται κανείς ότι θα χάσει τα κεκτημένα του και ούτε θα φοβάται κανείς ότι θα οδηγηθούμε σε έκρηξη λόγω της δυσπιστίας των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επόμενος ο κύριος Στάς για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Προεδρεύον. Μιλώ του πλέον ε, ξενόματος τη ομάδα μου και όχι ω εισηγητή για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια θα έχω την ευκαιρία επανέλθω. Να επαναλάβω μερικά πράγματα. Η ε, απαλλαγή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι μια ερώτηση και προ τον Επίτροπο αλλά και προ το Συμβούλιο. Η διαπίστωση ότι 80% των πόρων μας δαπανώνται από τα κράτη-μέλη και χρόνια ολόκληρα εδώ στο Κοινοβούλιο ζητούμε ε, δηλώσεις εθνικές για τη διαχείριση. Ο κύριος Λιμπεράς και όσοι συζητητής σε πολλές παραγράφους λέγει ότι θα πρέπει να υπάρχουν νέες ε, πλέον δυνατότητες, ε, νέα συνθήκη, άρθρο 317, νέες αρμοδιότητες και εξουσίες και υπάρχει δυνατότητα να κάνει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε το συντομότερο οι δηλώσεις αξιοπιστίας εθνικές να γίνουν υποχρεωτικές Κύριε ε, σε μετά το σκέφτεστε αυτό, ε, είστε διατεθειμένος να το δεχτείτε. Τέσσερα κράτη-μέλη το πράττουν ήδη, καλό είναι. Αλλά ε, με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους γίνεται αυτό. Ε, ας το συντονίσουμε λίγο, ας το τακτοποιήσουμε. το Συμβούλιο λέει τι κρίμα όμω υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που είναι ομοσπονδιακά κράτη, όπω το Βέλγιο, Βαλονία, Βρυξέλλες και ε, Φλάνδρα. Ε, και πώς μπορεί να έρθει με μια εθνική δήλωση αξιοπιστία. δεν είναι πρόβλημα αυτό αγαπητοί συνάδελφοι. Α, ας συμφωνήσει ως ε, εθνικός υπουργός με τους περιφερειακούς υπουργούς να περιμένει να συγκεντρώνει τις περιφερειακές εκθέσεις και το σύνολο μετά να το στέλνει στο κοινοβούλιο και στην κοινή γνώμη και να το δημοσιεύει και μπορεί να πει ότι μια χαρά ε, είναι η διαχείριση στις Βρυξέλλες και στη Βαλονία, στη Φλάνδρα Χάλια ή αντίστροφα, δεν ξέρω, ανάλογα. Ο κύριος ε, Λιμπεράτσκι επίσης ε, κάνει λόγο για την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την Προεταξιακή Βοήθεια προς την Τουρκία. Νομίζω ότι η διαπίστωση είναι λίγο ατυχής και ορισμένες παράγραφοι χρησιμοποιούνται με ε, κακό τρόπο και όχι παραγωγικό για την προενταξιακή διαδικασία και για τις διαπραγματεύσεις. Ο κύριος ε, Γκάιερ κάνει κάποιες προτάσεις, να το σκεφτείτε. Και τέλος προς το Συμβούλιο. Ελπίζω να μ' ακούτε κύριε Προεδρεύον. Θα μας απαντήσετε στη συνέχεια στην ερώτηση που σας έγινε μέχρι την 1η Ιουνίου 2010 να μας φέρετε αυτά που ζητάει το ψήφισμα στις παραγράφους 25-26. Θα μας απαντήσετε τώρα αν θα ανταποκριθείτε ή όχι σε αυτό το αίτημα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε ε, για να έχουμε κανονικές σχέσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στάς. Ακολουθεί κύριε Άσουορτ για δύο λεπτά. Ο κύριος Άσουορτ, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε λαμβάνω το λόγο ενώ του Βρετανικού Συντηρητικού Κόμματο και πάλι εφέτος θα καταψηφίσουμε την απαλλαγή του Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2008. Αυτή είναι μια πάγια στάση την οποία έχουμε ακολουθήσει με συνέπεια και θα εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτή τη στάση μέχρι ότου δούμε να υπάρχει μια πιο δυναμική αντιμετώπιση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το θετικό πιστοποιητικό ασφάλειας από το ελεγκτικό συνεδριό. Θέλω όμως να αναγνωρίσω δημόσια την πρόοδο η οποία έχει επιτελεστεί στη βελτίωση της, της δημοσιονομικής διαχείρισης από την προηγούμενη Κομισιόν. Το ελεγκτικό συνέδριο καταγράφει ιδιαίτερα την πρόοδο η οποία επετεύχθη στον τομέα της γεωργίας, της έρευνας, της ενέργειας, των μεταφορών και της παιδείας. Και θέλω να επενέσω την Κομισιόν για την πρόοδο που έχουν επιτύχει. Αυτό είναι ενθαρρυντικό το ότι υπήρξε αυτή η πρόοδος. Όμως, είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Πολλοί δρόμος παραμένει να τον διατρέξουμε. Το ελεκτικό συνέδριο και πάλι είχε αρνητικά σχόλια για την αδυναμία των ελέγχων, για πολλές ατασταλίες, για τον αργό ρυθμό ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβεβλημένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι παρά το γεγονός ότι η ευθύνη τελικά βρίσκεται στα χέρια της Κομισιόν, είναι τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο, ιδιαίτερα το Συμβούλιο που θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη ευσυνειδησία σε ό,τι αφορά την, ε, την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερες προσπάθειες για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το θετικό ΝΤΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, λειτουργούμε πια βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμεί το οφείλουμε στου Ευρωπαίους φορολογούμενου να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε στην κοινή γνώμη ότι πράγματι ο προπολογισμό δίνει προστιθέμενη αξία με τα χρήματα τα δημόσια και ότι υπάρχει μια ακαιρεότητα στις εσωτερικές οριστικές διαδικασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι ότου δοθεί το θετικό DAS από το ελεκτικό συνέδριο, εγώ και το κόμμα μου θα εξακολουθούμε να καταψηφίζουμε τις απαλλαγές του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άσουεθ για πέντε λεπτά ο κύριος Ζόντεργαρντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η συζήτηση που κάνουμε αφορά το να διαπιστώσουμε αν ως ευρωβουλευτές, ο καθένας ατομικά και συνολικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι καλώς έγινε η διαχείριση του προϋπολογισμού του 2008. Γιατί ούτως ή άλλως ε, όταν φτάσει ο μήνας Μάιος, εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Η ομάδα μου έχει ε, ένα πολύ επικριτικό, μια πολύ επικριτική θέση και στάση απέναντι ε, στο θέμα αυτό. Σε ορισμένους τομείς όντως υπήρξε πρόοδο σε σχέση με το 2007, αλλά υπάρχουν πολλοί άριθμοι τομείς επί των οποίων τα αποτελέσματα είναι ανεπαρκή. Παραδείγματος χάρη λογαριασμοί της ε, Κομισιόν. Το... Και τα διαφορετικά... Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι το 11% των κονδυλίων πληρώθηκαν με βάση τους κανόνες. Και για λόγους λαθών και για λόγους απάτης. Το αποτέλεσμα ποιο είναι ότι δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτό το τομέα δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί και παρόλα αυτά κατεβλήθησαν. Αυτό είναι δεκτό και παραδεκτό. Γνωρίζουμε όλες τις δικαιολογίε. Η Κομισιόν ρίχνει τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη, γιατί εκείνα είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο. Τα κράτη-μέλη λένε ότι είναι υπεύθυνη η Κομισιόν, γιατί οι κανόνε είναι πάρα πολύ περίπλοκοι. Είναι πολύ εύκολο να παίζουμε αυτό, πινκ-πονγκ, μεταξύ οργάνων. Το θέμα που τίθεται όμω είναι αν επρόκειτο για ένα ίδρυμα, για, ένα ποδοσφαιρικό, για μια ποδοσφαιρική ομάδα, για ένα πολιτικό κόμμα. Και αν ένα τόσο σημαντικό τμήμα των κονδυλίων είχαν καταβληθεί με αυτόν τον τρόπο, θα δεχόμασταν τους λογαριασμούς. Εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνουν διαφορετικές αλλαγές. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Η διαδικασία της απαλλαγής, λοιπόν, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υπάρξει αλλαγή για να πιέσουμε το Συμβούλιο. Πέρυσι τον Απρίλιο το Κοινοβούλιο αρνήθηκε την απαλλαγή για τους λογαριασμούς του Συμβουλίου το 2000, για το 2007. Είχαμε πει πέρυσι ότι δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο δεν δεσμευόταν να μας συναντήσει. Να συναντήσει την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να απαντήσει τις ερωτήσεις της. Εμείς θέλησαμε να δείξουμε καλή θέληση και τον Νοέμβριο παρόλα αυτά δώσαμε την απαλλαγή στο Συμβούλιο. Αλλά θέσαμε κάποιους όρους και κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες ήταν ξεκάθαρες. Απαιτήσαμε να υπάρξει αλλαγή από φέτος. Παρόλα αυτά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ούτε μία αλλαγή έχει συμβεί. Να σας δώσω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μάλιστα. Το Συμβούλιο μεταφέρει δισεκατομμύρια ε, ευρώ από λογαριασμό σε λογαριασμό. Γιατί θα κάνει αυτό το Συμβούλιο, γιατί κάνει αυτές τις ε, μεταβιβάσεις. το χάρη τεράστια ποσά που τα μεταφέρει στο λογαριασμό για τα ταξίδια. Ποιος τα χρησιμοποιεί αυτά τα λεφτά. Άτυπα το Συμβούλιο μας απαντάει, αλλά ποτέ δεν έχει δεχθεί να μας απαντήσει σοβαρά, επίσημα και δημόσια. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να χορηγήσουμε την απαλλαγή στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να δεσμευτεί το Συμβούλιο, να απαντήσει στις ερωτήσεις μας, να δείξει διαφάνεια και καλή θέληση απέναντι στο Κοινοβούλιο οι κριτικές μας απέναντι στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν είναι ξεκάθαρες. Και πολλοί άλλοι συναδέλφοι από άλλες ομάδες συμφωνούν μαζί μας. Αλλά ακριβώ ε, γι' αυτό πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας για τη δική μας οικονομική διαχείριση, για τους λογαριασμούς δηλαδή του Κοινοβουλίου Γι' αυτό ακριβώ είμαστε δυσαρεστημένοι πραγματικά, που η έκθεση που μας αφορά είναι λιγότερο επικριτική, λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επανισάγουμε κάποιες κριτικές σε αυτή την έκθεση. Κάποια πιο αυστηρά σημεία και σχόλια. Η αυτοκριτική θα μας δώσει το Μάιο μεγαλύτερη δύναμη και θα καταστήσει την κριτική μας πολύ πιο δρυμία απέναντι στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Οι συνάδελφοι της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού φέτος θα ήθελα να δείξουν μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στα χρήματα του καταναλωτή. Του φορολογούμενου, συγγνώμη. Ευχαριστώ η κυρία Ανδρέα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Αγαπητοί συνάδελφοι, η, η απαλλαγή είναι η πιο σημαντική πράξη για την οποία ευθυνόμαστε. Πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε, να ελέγξουμε πώς ξοδεύονται τα χρήματα των ε, Ευρωπαίων ε, φορολογουμένων και να παρακολουθήσουμε ε, την ε, τον έλεγχο των ε, δαπανών. Βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν ορισμένες δαπάνες οι οποίες δεν αιτιολογούνται παρκώς. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί απαλλαγή βάσει στην βελτίωση της χρήσεως των ευρωπαϊκών πόρων. Πρέπει όμως να σας πω ότι αυτό που θέλουν να ξέρουν οι φορολογούμενοι είναι αν τα χρήματα δόθησαν στα κατάλληλα άτομα και ε, σε σωστό ύψος. Οπότε, ε, εφόσον ε, περί αυτού πρόκειται η απαλλαγή, τα τελευταία χρόνια η μόνη βελτίωση από την Επιτροπή το Συμβούλιο και το Συμβούλιο είναι μετατοπίσεις μεταξύ κρατών μελών. Αλλά το θεσμικό όργανο στο οποίο αναθέτει τη διαχείριση των χρημάτων ο Ευρωπαίος Χορολογούμενος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή λοιπόν θα έπρεπε να προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους προτού ε, ε, ε, διαθέσει τα χρήματα. Ε, υπάρχει βέβαια ένα ανεκτό ποσοστό λαθών. Γιατί πρέπει κανείς ε, να ε, επιτρέπει ένα ανεκτό ποσοστό αταξίας εφόσον θα πρέπει να υπάρχει απολογισμός. Πέρυσι καθυστέρησε μέχρι τον Νοέμβριο η απαλλαγή και παρόλο που δεν έγινε δεν διεξήχθη κριτική κατά της διαχειρήσεως. Εφέτος εμείς απευθυνόμαστε στο Συμβούλιο και προτείνουμε να καθυστερήσουμε. Είμαστε όμως σοβαροί για τις ευθύνες μας ή κάνουμε πολιτικά παιχνίδια εδώ. Πρόκειται για ένα διαθεσμικό παιχνίδι ε, όταν μιλάμε για την απαλλαγή. Ε, μπορούν να το ανεχτούν πλέον οι φορολογούμενοι εφόσον δικά τους είναι τα χρήματα. Παρακαλώ λοιπόν λοιπόν όλοι να εξασκήσετε τις ευθύνες σας πολύ προσεκτικά και να ε, ε, ε, ζητήσετε να μην υπάρξει απαλλαγή για κανένα από τα θεσμικά όργανα τα οποία δεν προασπίζουν τα συμφέροντά μας μέχρι ότου να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει χρηστή διαχείριση. Ευχαριστώ κυρία Ανδρέασεν επί διαδικοστικού ο κύριος Δανέσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, διότι βλέπω το όνομα Λόπες Γκαρίντο δηλαδή δόξα το Θεώ υπάρχει κάποιος ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Συμβούλιο θα αναφερθεί όμως και σε αυτά τα οποία είπα εγώ σχετικά με τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου και την ε, έλλειψη ε, χρηστής εκτελέσεως αυτού του προπολογισμού εφόσον δεν με άκουσε, εφόσον τώρα μόλις έφτασε, καθυστέρησε δηλαδή. Ε, είπατε ότι ζητάτε κάτι διαδικαστικό. Έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, να κάνετε κάποια πρόταση σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στον Υπουργό να απαντήσει στην ερώτησή μου, άρα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπα στην αρχή. Ε, μου είπατε ότι ο κύριος Γκαρίντο είναι στην, ε, ε, στο κατάλογο των ομιλητών, είναι όμως ελεύθερος και θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Έρενχάουζερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε ένα σημείο συμφωνούν όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Χρειαζόμαστε ε, μία λύση για το σύστημα των ευρωπαϊκών οργανισμών και έχω να κάνω μία πρόταση κατά τρόπο να ε, εξοικονομούμε ετησίως μισό δισεκατομμύριο ευρώ χωρίς ε, να μειωθεί η αποδοτικότητα των προγραμμάτων. Πρώτον, να υπάρχει μία καλύτερη πρωταρχική βάση η οποία δεν δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της Λισαβόνους. Δεύτερον, να υπάρχει μία αξιολόγηση της προστιθεμένης αξίας προτού διατεθούν οι πόροι. Ε, τρίτον, ε, ε, ενδελεχής έλεγχος όλων των μεμονωμένων δαπανών. Τρίτον, όλα αυτά να είναι υπό την ευθύνη ενός μοναδικού επιτρόπου που θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση AUTHORWAVE ε, μείωση των μελών των ε, διαχειριστικών ε, συμβουλίων, διοικητικών συμβουλίων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος κριτηρίων όπως ανέφεραν προλαλήσαντες. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των πολιτών. Στα γραφεία αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ανεξάρτητο καθεστώς και αφού εισακουστεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνενέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, επιλεγεί ε, ε, μία πορεία. Θα πρέπει να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της Επιτροπής και των οργανισμών αυτών βάσει κριτηρίων που θα καταρτίζει το ελεγκτικό συνέδριο. Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία τράπεζα δεδομένων κατά τρόπον εμείς να κάνουμε στατιστικές αξιολογήσεις που δεν δεν μπορούμε να, μπορούμε να κάνουμε τώρα διότι λαμβάνουμε όλα τα έγγραφα μόνο σε χαρτί ε, και όχι σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης ε, υπάρχουν λύσεις. Ε, είναι προφανές. Θα έλεγα λοιπόν να επιτρέψετε να εφαρμοστούν οι λύσεις αυτές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Έρεν Χάουζερ και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Λόπες Γκαρίντο για το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι ενώπιόν σας. Παρότι δεν με είχατε προσκαλέσει επίσημα, δεν με είχε προσκαλέσει επίσημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παραστώ σε αυτή τη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, όταν έμαθα ότι υπήρχε ένα αίτημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από κάποιους ευρωβουλευτές για να παραστώ, αμέσως, με τα χαράς, ήρθα για να παραστώ σε αυτή τη συζήτηση. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου που αφορά το έτος 2008 ήταν σωστή, ορθή και αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Έγινε μια παρέμβαση από τον κύριο Σόντεγκάρντ που μίλησε για διαφάνεια. Για απουσία, μάλιστα, διαφάνειας. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και θα είμαι ξεκάθαρος. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι με απόλυτα διαφανή τρόπο εκτελεί τον προϋπολογισμό του. στο βαθμό που εκτελεί ορθά τον προϋπολογισμό με βάση όλες τις ε, προϋποθέσεις για την εκτέλεσή του. Επιπλέον, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο στην ιστοσελίδα του δημοσιεύει μια έκθεση για την ε, δημοσιονομική διαχείριση του προηγούμενου έτους. Θα ήθελα επίσης να σας ε, επιστήσω την προσοχή σε αυτό να σε πείσω προσοχή στο γεγονός ότι σήμερα το Συμβούλιο είναι το μοναδικό όργανο που έχει δημοσιεύσει μια έκθεση προκαταρτική για τους λογαριασμούς του 2009, για το κοινό εν γέννη, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, πριν από λίγες μέρες, στις 15 Μαρτίου, ο πρόεδρος του Κορεπέρ και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συναντήθηκαν με μια αντιπροσωπεία της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Και κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού του Συμβουλίου του 2008. Ο κύριος Γερμπράντι έκανε μία ερώτηση για την ανάγκη βελτίωσης και εξέλιξης. Είπε ότι θα αμοιβαίως έλεγχος χωρίς συμφωνία κυρίων. Πρέπει να ξεπεράσουμε, είπε, τη συμφωνία κυρίων. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να αναθεωρηθεί αυτή η συμφωνία, το Συμβούλιο είναι στη διάθεσή σας για να το εξετάσει, να το συζητήσει, για να υπάρξει ενδεχομένως μια νέα συμφωνία που να βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Και αν χρειαστεί να φτάσουμε σε νέα συμφωνία καλύτερη ή δυνατόν από τη σημερινή. Αυτά ήθελα να πει το Συμβούλιο για τη συζήτηση που έγινε σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση που μου απευθύνατε. Θέλω να επαναλάβω ότι εγώ δεν είχα ενημερωθεί επίσημα για το γεγονός αυτό, όλα αυτά ήρθα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, Σα ευχαριστούμε για το γεγονό ότι ανταποκριθήκατε στην επιθυμία του Κοινοβουλίου. Βέβαια, ούτε για την Κομισιόν, ούτε για το Συμβούλιο υπάρχει μια επίσημη πρόσκληση που πρέπει να απευθύνεται για να είναι παρούσα και εδώ όπως και εσείς. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο πάντα θα πρέπει να είναι παρόν στις συνεδριάσεις μας, ιδίως οι εκπρόσωποι της Προεδρίας. Ο κύριος Σοντή έχει τώρα το λόγο, είναι ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Σεμέτα, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και οι πρώτες μου λέξεις θα είναι τα ευχαριστήρια Προ τον Μπογκουσλάβ Λιμπεράσκι, ομιλώ εξ τη της ομάδας του ΕΛΚ, σε σχέση με την απαλλαγή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτο 2008. Θέλω να ευχαριστήσω και του συνεισηγητέ από τα άλλα πολιτικά κόμματα και τον κύριο Καλντέιρα από το Ελεκτικό Συνέδριο, ο οποίο έχει κάνει μαζί με τι υπηρεσίε του μια τεράστια εργασία για να μπορέσει να μα διαφωτίσει αυτέ τι πολυδέδαλε διαδικασίε. Η ομάδα μου υποστήριξε την ε, απαλλαγή της Επιτροπής στην αρμόδια Επιτροπή κυρία Σεμετά και εμείς διαπιστώνουμε ότι υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι χάρη στην εργασία και του προκατόχου σας του κυρίου Σιμ Κάλλας. Αλλά σε ό,τι αφορά τους ετήσιου λογαριασμού καταρχήν, η δήλωση του ελεκτικού συνεδρίου είναι θετική. Δίνει το θετικό πιστοποιητικό αξιοπιστίας. Ίσως λοιπόν κάποτε και οι συντηρητικοί κύριοι Άσχουρθ θα δεχτούν να ψηφίσουν τουλάχιστον θετικά για τους ετήσιους λογαριασμούς. Αλλά εξακολουθώ να έχω ανησυχίες για το γεγονός ότι έχουμε αρνητικού ίδιους πόρους 50 εκατομμύριων ευρώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν καταγράφουμε τις ε, υποχρεώσεις έναντι των κρατών μελών που είναι ακριβώς τα ποσά που έχουν να κάνουν με τη συμβολή τους στα, στις συντάξεις των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουμε αρνητικό πιστοποιητικό σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 287 για το ζήτημα αυτό που αφορά πράξεις οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία αυτή. Έχουμε τη γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου που καλύπτει πέντε παραγράφους, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς προτείνεται. Τι ακριβώ αναφέρει το ελεκτικό συνέδριο, θα θέλαμε να ξέρουμε στην περίπτωση αυτή αν οι αποστολέ αυτέ του Συμβουλίου εγγρα... εγγράφονται μέσα σε αυτά τα οποία ζητά η συνθήκη για τη μεθοδολογία. Ζητούμε από τις κυβερνήσει μας να έχουμε δηλώσει αξιοπιστίας που δεν παίρνουμε ποτέ από τα εθνικά κράτη. Γι' αυτό εγώ προτείνω τα εθνικά λογιστικά όργανα, τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια να συμμετέχουν στην αλυσίδα πιστοποίηση, να δίνουν πιστοποιητικά εξ ονόματος των κυβερνησεών του. Πρέπει να μειωθεί ο χρονικός ορίζοντας για την απαλλαγή. Είναι 2012 σήμερα και εμείς μιλάμε ακόμα για, για την απαλλαγή του 2008. Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία να καθυστερήσουμε να εγκρίνουμε την απαλλαγή του Συμβουλίου, γιατί το ελεκτικό συνέδριο δεν έκανε καμία απολύτω παρατήρηση στον τομέα αυτό. Εγώ προτείνω μια να καθυστερησουμε να εγκρινουμε την απαλλαγη του συμβουλιου γιατι το Ελεκτρικό συνεδριο δεν συνδιάσκεψη με Συμβούλιο, Κομισιόν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Εθνικών ελεκτικό συνεδρίων για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία απαλλαγή και να μπορέσουμε να διαλευκάνουμε όλα αυτά τα ιδίως, ιδιαίτερα τεχνικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Όντι. Η κυρία Βάιλερ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ εκπρόσωπε της Κομισιόν και επίσης και του Συμβουλίου. Κάθε χρόνο έχουμε αυτή τη συζήτηση για, τη... για βελτιώσεις ή στην ε, ε, διαχείριση των ε, ευρωπαϊκών πόρων για καλύτερους ελέγχους, για μεγαλύτερη διαφάνεια για το Κοινοβούλιο και τους πολίτες. Η πρώτη ένδειξη είναι ήδη η παρουσία του Συμβουλίου, ότι κάτι αλλάζει και στο Συμβούλιο. Χαίρομαι πολύ που το καταλάβατε, αλλά δεν επαρκεί, διότι εσείς είστε της γνώμης ότι έχετε αποκαταστήσει πλήρη διαφάνεια και νομίζετε ότι οι ερωτήσεις ε, ε, ε, εάν όμως λάβετε υπόψη σας ότι οι ερωτήσεις του Νοεμβρίου ακόμη δεν έχουν λάβει απάντηση υπάρχει μια μεγάλη διάσταση απόψεων και θα πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα διότι θέλετε να δημιουργήσετε νέα βάση επεξεργασίας αλλά η προσμονή μας δεν είναι νέα είναι κάτι το οποίο έχουμε απαιτήσει επανειλημμένως και τώρα το συζητάτε σαν να είναι ε, κάτι που προκύπτει για πρώτη φορά. Ε, συμφωνούμε με την κριτική των ε, διαφόρων πολιτικών ομάδων. Δεν θα απαλλάξουμε το Συμβούλιο ούτε αυτό το μήνα ούτε τον επόμενο. Και όπως είπε και η κυρία Ανδρέας, συμφωνώ ότι ναι, εφόσον μεν τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για 80% της διαχειρίσεως των χρημάτων δεν απαλλάσσεται το Συμβούλιο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε. Χρειάζεται όμως συγχρόνως και συνέπεια. Πρέπει να βελτιώσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε διότι κάθε χρόνο σηκώνουμε την κίτρινη κάρτα της μη απαλλαγή και δεν συμβαίνει τίποτα. Άρα δεν επαρκεί κριτική αλλά πρέπει κανείς να τονίσει και τις επιπτώσεις του τι μέλη γενέστε αν το Συμβούλιο δεν συνεργάζεται σωστά, δηλαδή θα χρειαστούν νέες θεσμικές αλλαγές. Ευχαριστώ κυρία Βάιλερ. Κυρίες και κύριοι, ε, τώρα μόλις ε, ε, επαλήθευσα εις, την, στον εσωτερικό κανονισμό. Ε, θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι δικαιούμαστε να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Χατζημαρκάκη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του και έχει λόγο για μισή λεφτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, κύριε Επίτροπε Σεμέτα, ε, ένα από τα βασικά καθήκοντα είναι, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η χορήγηση απαλλαγής και η διαχείριση των χημάτων είναι ένα βασικό θέμα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω καταρχήν για τις εκθέσεις αλλά βλέπω και φως και σκύρα Δηλαδή φως υπάρχει όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει και διαχειρίζεται μόνη της τα χρήματα. Αλλά αν αυτό είναι αποτελεσματικό είναι κάτι τελείω διαφορετικό και πρέπει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να απασχοληθούμε περισσότερο με την αποτελεσματικότητα και ιδίω να τονίσουμε περισσότερο τις προοπτικές ε, της Ατζέντα 2020 διότι υπάρχει, υπάρχουν σκιώδεις τις περιοχές ε, όπου ε, υπάρχουν ε, πόροι οι οποίοι έχουν διατεθεί λανθασμένα και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει 100% αυτών των χρημάτων να επιστραφούν. Δεν είναι εύκολο να απαλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι υπήρξε καθυστέρηση της εφαρμογής συνθήκης της Λισαβόνας και ίσως πρέπει να κοιτάξουμε αν όλα αυτά δεν έχουν οδηγήσει σε περισσότερη συγκάλυψη των ε, συνθήκων ε, διότι υπάρχει κατανομή των ε, αρμοδιοτήτων των επιτρόπων και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ελέγξουμε. Όσον αφορά όμως τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τη Συμφωνία Κυρίων έχω να πω ότι μεταξύ 2008 και 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε πάνω από 300 εκατομμύρια στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για αναπτυξιακή βοήθεια αλλά και ε, ε, για ε, οργανισμούς οι οποίοι προσπαθούν να καταστρέψουν την, το κύρος Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν κατάλογο και μία αξιολόγηση όλων αυτών των αποδεκτών Όσον αφορά τον κύριο εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ και θα να του πω ότι επεξεργαζόμαστε ε, πολλά χρόνια τώρα τη Συμφωνία Κυρίων, κυρίων ε, ε, χρειάζεται να προωθηθεί και η συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χατζημαρκάκη. Η κυρία Φόξ για δύο λεπτά έχει το λόγο τώρα. After the Fox. Ευχαριστώ. Fox. Πάλι μας ζητάτε να δώσουμε απαλλαγή ε, ενός σημαντικού αριθμού λογαριασμών. Μιλάμε για λογαριασμούς όπου το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει δώσει θετική δήλωση αξιοπιστίας ε, και που δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι νόμιμοι και εντάξει. Οι ελεγκτές είπαν ότι υπάρχουν σωρία παρατυπιών στους λογαριασμού και παρόλα αυτά πρέπει να του επικυρώσουμε εμεί. Χαίρομαι που η κυρία Ματιό σύστησε την αναβολή της απαλλαγής για την Ευρωπαϊκή, Ακαδημία Αστυνομία, Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να διερευνήσουμε τους λογαριασμούς. Επίσης υπάρχουν ισχυρισμοί ότι υπάρχουν πολλές απάντες σε αυτήν την Ακαδημία ε, και θεωρείται ότι το προσωπικό χρησιμοποιεί λεφτά ε, για να αγοράσει δικά του έπιπλα. Ε, δεν δεχόμαστε αυτές τις παρατυπίες. Θα πρέπει να αρνηθούμε την απαλλαγή μέχρι το ελεκτικό συνέδριο δώσει θετική δήλωση αξιοπιστίας. Η εμπιστοσύνη στην πολιτική ε, έχει βυθιστεί. Και νομίζω ότι εμείς ε, θα χειροτερέψουμε τα πράγματα εάν επικροτήσουμε τέτοιες πατάλες. Κάθε φορά που απαλλάσσουμε τέτοιους λογαριασμούς ενθαρρύνουμε την απάτη και τη σπατάλη. Κάθε φορά στέλνουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο, στην Κομισιόν και στους φορολογούμενούς μας ότι δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό σοβαρά. Το κόμμα μου θα εξετάσει πολύ προσεκτικά πώς οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές βουλευτές αποφασίζουν να χειριστούν αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε την πολιτική, να υπάρξει εκαθάριση και παρόλα αυτά κάθε χρονιά να δεχόμαστε τέτοιους λογαριασμούς. Οποιοδήποτε είναι σοβαρό και πραγματικά θέλει τη μεταρρύθμιση, πραγματικά θέλει να προστατεύσει τα λεφτά των φορολογούμενων, θα πρέπει να αρνηθεί την απαλλαγή. Ευχαριστώ κύριε Φόξ. Για ένα λεπτό κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή είναι υψηλό το ποσοστό των ατασταλιών και των ελλείψεων, εγώ είμαι αρνητικό σε σχέση με το θέμα τη ε, απαλλαγή για την Κομισιόν. Θα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερο για την ε, απλοποίηση των κανόνων, ιδίω σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία. υπήρξαν πολλοί ανεξάρτητοι φορεί οι οποίοι έκαναν προτάσει σχετικά, αλλά η Κομισιόν δεν έχει απαντήσει σε αυτά. Μια ανεξάρτητη εξωτερική έρευνα για τα θέματα αυτά είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει. Και επομένω θα πρέπει η υψηλή ψηλού επίπεδο ομάδα υπό τον κύριο Στόιμπερ να επιληφθεί του θέματος αυτού. Θα πρέπει επομένως να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η σωστή υποστήριξη για αυτές τις ενέργειες. Για μας δεν είναι μονάχα θέμα της μείωσης και της συμπίεσης του διοικητικού κόστους, αλλά πολύ περισσότερο να εξασφαλίσουμε το κόστος εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών θα είναι μικρότερο. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε να περάσει από τα χέρια μας αυτή η ευθύνη. Χρειαζόμαστε να υπάρξει καλύτερη διαλεύκανση πολλών στοιχείων και να μειώσουμε και το άχθος της διοίκησης για τρία λεπτά ο κύριος Χόλμα, η κυρία Χολμάερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στα προβλήματα της αναψυξιακής βοήθειας που μας υποδεικνύονται από το ελεγκτικό συνέδριο. Και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιάλα Σέντερ για την καλή συνεργασία με την οποία αντιμετωπίσαμε τα θέματα αυτά. Πρώτα απ' όλα, τίθεται η προβληματική της ε, βοήθειας σε επίπεδο προϋπολογισμού των αναπτυσσόμενων χωρών, η οποία όμως υπόκειται πάντα στην υποψία ότι βοηθάμε διεφθαρμένα και ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα οποία καταπιέζουν του πληθυσμού τους και δεν δίδεται καμία πραγματική βοήθεια σε αυτές τις ομάδες. Και πολλές φορές υπάρχουν <coughs> πολλές κριτικές απόψεις για τα θέματα αυτά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να μειωθούν ή ακόμα και να καταρριχθούν τελείως για τις χώρες όπου υπάρχει πραγματικά ε, ύπαρξη προβλημάτων σε σχέση με τη χρήση αυτών των επιδοτήσεων σε επίπεδο προϋπολογισμού. Επίσης είναι διάτριτες αποσφάλματα οι οι λογαριασμοί, οι λογαριασμοί για την ε, βοήθεια που δίνονται σε διάφορους φορείς και δεν υπάρχουν πολλές φορές ούτε θεσπίσεις σαφών προτεραιοτήτων. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι ακριβώς αποσκοπούν αυτά τα κονδύλια για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα των σχεδίων που αφορούν τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αποδειχθούν πράγματι προς το όφελος του τοπικού πληθυσμού. Η αναπτυξιακή βοήθεια λοιπόν γενικά θα πρέπει να ενσωματωθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη συγκεκριμένα στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχομαι τώρα στο θέμα τη Τουρκία. Εγώ εξεπλάγει για το γεγονό ότι απόλυτα φυσιολογικέ κριτικέ, οι οποίε εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιούνται για άλλε χώρε σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων, στην περίπτωση τη Τουρκία υπήρξε κατά κάποιο τρόπο μια απόλυτη παράκαμψη αυτών των προβλημάτων. Θα πρέπει να γίνεται ο καθορισμός των στόχων και των κατευθύνσεων των σχέδων από την πλευρά της Κομισιόν, αλλά η Κομισιόν θα πρέπει στη συνέχεια να εξασφαλίζει ότι έχουν πράγματι εκτελεστεί τα προγράμματα αυτά με σωστό τρόπο. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων, θα πρέπει να το υποδεικνύει αυτό η Κομισιόν και να το αναφέρει. Και εδώ ξέρω ότι ένα μέρος των ε, προγραμμάτων δεν έχει εκτελεστεί σωστά και γι' αυτό προτείνουμε να υπάρξει μια παρακράτηση, μια ε, ένα πάγωμα ενός ορισμένου αριθμού των ποσών, ώσπου να μπορέσουν πραγματικά να εκτελεστούν σωστά αυτά τα σχέδια. Υπήρξαν αντίστοιχε επικρίσει για χώρε όπω η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ελλάδα και μια τέτοια διαδικασία ακολουθήθηκε σε αυτήν την περίπτωση. Επίση, σε ό,τι αφορά την κτηριακή πολιτική, νομίζω ότι θα πρέπει να έχει ένα σαφή σχεδιασμό σε μικροσοπρόθεσμο επίπεδο αυτή η πολιτική και θα είναι απαραίτητο με τον τρόπο αυτό να μην πληρώνουμε πρόσθετο, πρόσθετα κονδύλια για ενδιάμεση χρηματοδότηση. Θα πρέπει η πολιτική αυτή να είναι σαφής και να μπορέσει να σχεδιαστεί με έναν τρόπο που θα είναι απόλυτα Σε Ένα τελευταίο σημείο κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη απλοποίηση και έλλειψη πολυπλοκότητος σε πάρα πολλά σχέδια και προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι μόνο μια ρητορική διεκδίκηση, είναι κάτι το οποίο πρέπει επιτέλου να εφαρμοστεί και στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Χολμάιερ. Ακολουθεί ο κύριος Γκάιερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Γενικέ Γραμμάτε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που βρίσκετε εδώ και έτσι τονίζετε τη σημασία της συζητήσεώς μας. Ε, ξέρετε ε, τα τεχνάσματα. Ε, αν θέλετε να φέρετε κάποιον σε δύσκολη θέση, κάντε μία ερώτηση. Του λέγεται χτυπάτε ακόμη, δέρνετε ακόμη τα παιδιά σας. Αν σας πει όχι, σημαίνει ότι το έχει κάνει στο παρελθόν. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη συνεργασία. Ο συνάδελφος Στάς έχει κάνει μία κατακριτική έκθεση και σε ορισμένα σημεία ακολούθησε αυτού του είδους την λογική και ε, ε, πρέπει να υπάρχει η ε, κριτική αλλά πρέπει να είναι σωστή. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να απορριφθούν ορισμένες απόψεις που διατυπώνονται στις εκθέσεις αυτής απαλλαγής και θέλω να απαριθμίσω εδώ αυτά που με απασχολούν διότι αναφέρονται ή στην πραγματικότητα και δεν εφαρμόζονται εφαρμόζονται ή που δεν βοηθούν το να δημιουργήσουμε νέες αρχές μεταξύ της Προεδρίας και της Ολομελίας και υπάρχουν και καλές προτάσεις οι οποίες έχουν υιοθετηθεί. Αλλά εδώ καλύπτουμε μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας όπως την τροπολογία 26 η οποία ζητά την εφαρμογή ενός εσωτερικού ελεγκτικού συστήματος από τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου αλλά στην σοσιαλιστική ομάδα αυτό έχει όντως υλοποιηθεί παρόλο που πιστεύουμε ότι χρειάζονται ακόμη προσπάθειες και μπορούμε να συμφωνήσουμε μόνο εάν παρουσιάσει κανείς την πραγματική κατάσταση στην έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσουμε μία διατύπωση η οποία να λέγει ότι όντως αυτό είναι γεγονός ή στη σοσιαλιστική ομάδα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάγερ, ο κύριο Σμιτ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Sorry. Γινόμαστε όλο και καλύτεροι στον έλεγχο του προπολογισμού. Και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Δεν πρέπει να σπαταλιέται ούτε ένα σέντ για το Αναπτυξιακό Ταμείο. Εμείς είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής, η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ. Και αυτό είναι καλό. Είναι καλό να δείχνουμε αλληλεγγύη με τους στοχότερους ε, σε αυτόν τον κόσμο αλλά νομίζω ότι παρότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θέλουν να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες, τα χρήματα αυτά θα πρέπει να ε, χορηγούνται ε, με τρόπο ε, συνετό. Δεν θα πρέπει να τα δίνουμε σε διεφθαρμένους ηγέτες. Δεν θα πρέπει τα χρήματα αυτά να μην δίνουν αποτελέσματα, να μην χτίσουν το μέλλον. Και εδώ το Κοινοβούλιο έχει τεράστια ευθύνη. Οι διάφορε επιτροπέ έχουν υποβάλει τροπολογίε και οι συγητές ήταν πολύ θετικοί απέναντι σε αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαιτήσει από αυτέ τι χώρες που τι υποστηρίζει να πληρούν και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραδείγματο χάρη ελευθεροτυπία και ελευθερία έκφραση. Δυστυχώ αυτό δεν συμβαίνει παντού σήμερα. Να σα δώσω ένα σαφέ παράδειγμα. Εμεί ε, υποστηρίζουμε την Ερυθρέα. Στην Ερυθρέα Όσοι επικρίνουν την κυβέρνηση φυλακίζονται χωρίς καμία δίκη και χωρίς να έχουν κατηγορηθεί και για τίποτα μάλιστα. Επί χρόνια σαπίζουν στη φυλακή σε φρικόδεις συνθήκες. Εμείς τι κάναμε για να επικρίνουμε την ε, κυβέρνηση και τον πρόεδρο της χώρας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασκήσουμε ξεκάθαρες κριτικές. Όταν οι χώρες δεν σέβονται τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να μπορούμε να ακυρώνουμε την υποστήριξή μας προς αυτές τις χώρες. Και ζητώ από το Συμβούλιο να με ακούσει πάρα πολύ προσεκτικά. Ε, νομίζω ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να εκφράζει τέτοιες απόψεις. Αυτό περιμένουν από μας οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Σμίτο. Κύριος Φαντάλεν, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κυρίου Στάς έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία αφορούν πολύ σημαντικά θέματα. Όλοι εμείς είμαστε δημόσια πρόσωπα και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες ανα πάσα στιγμή. Θα πρέπει να δείχνουμε ανα πάσα στιγμή στους πολίτες που το επιθυμούν α, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε ε, και το τελευταίο ΣΕΝΤ το Κοινοβούλιο τα προηγούμενα χρόνια ε, βελτιώθηκαν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν θέματα με τα έξοδα των ε, βουλευτών. Κάθε χρόνο θα πρέπει εγώ, παραδείγματος χάρη, να, να προσλαμβάνω ένα λογιστή για να ετοιμάζω τα τους λογαριασμούς μου. Γι' αυτό η τροπολογία 33 είναι πάρα πολύ σωστή. Αφορά την ε, παράγραφο 65 της έκθεσης αυτής. Είναι πολύ σημαντική Αν την υποστηρίξετε παρακαλώ. Κυρία Γιαρτσεβέσκα για 1,5... Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το γραφείο έψω για την πρόσληψη προσωπικού είναι ο φορέας ο οποίος εξασφαλίζει τη στελέχωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Χαίρομαι που η έκθεση απαλλαγής αναφέρεται και σε αυτό το σημείο. Πρέπει να καταβάλουμε τις κατάλληλες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πραγματικά θα υπάρχουν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους υποψήφιους για να γίνουν μέλη του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν έχουμε πάρα πολύ λίγους υπαλλήλους από τα νέα κρατημέλη, κατά την άποψή μου, εάν λάβουμε υπόψη την κατάσταση του των ανωτέρων στελεχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελάχιστη η υπάλληλοι από τα κράτη-μέλη της ε, Ανατολικής Ευρώπης. Είναι μακρά η διαδικασία για την πρόληψη, πρόσληψη, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν επιτύχει στους διαγωνισμούς, πολλές φορές πρέπει να περιμένουν τόσο πολύ ώστε προτιμούν να πάρουν άλλες θέσεις εργασίας, ώστε εφόσον δεν βλέπουν να τελειώνει αυτή η διαδικασία σε επίπεδο έψω. Υπάρχει ένα σχέδιο μεταρρύθμισης για την ε, διαδικασία στελέχωσης και η έψω έχει αναγνωρίσει και ορισμένες από τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ θα παρακολουθήσω λοιπόν την πρόοδο αυτού του εγχειρήματο ε, μεταρρύθμισης και θέλω να τονίσω ότι το έψο θα πρέπει να προσελκύσει τους καλύτερους στην αφρόκρεμα για να έχει τους καλύτερους υποψηφίους και να εξασφαλίσει ότι θα έχουμε τους, καταλή, τους καλύτερους καταλόγους επιτυχόντων, οι οποίοι όμως να εκφράσουν και τη γεωγραφική κατανομή των υποψηφίων μεταξύ των 100 μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ο κύριος Κάλφιν για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας μιλήσω για την απαλλαγή των εκτελεστικών ε, υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου κυρίου Σταυρακάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, παρότι εκ μέρους των σοσιαλιστών ήταν ο εισηγητής και συνεισηγητής και δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είχε πρόβλημα με τις μεταφορές. Σε ό,τι αφορά την ε, ορθή χρήση του προϋπολογισμού των εκτελεστικών υπηρεσιών, των εκτελεστικών agencies, αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια την κυρία Ματιέ, καθώς και τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου και τους υπευθύνου των ε, ε, υπηρεσιών αυτών με τους οποίους συνεργαστήκαμε. Θα ήθελα να σας πω ότι ο προϋπολογισμός αυτών των υπηρεσιών είναι μια διαδικασία και ο έλεγχός της είναι πάρα πολύ επαχθή διαδικασία, διότι η εκτέλεση γίνεται με τελείω διαφορετικό τρόπο από υπηρεσία σε υπηρεσία. Βεβαίω, η εκτέλεση του προπολογισμού βελτιώνεται από χρόνο σε χρόνο. Και οι υπηρεσίε δέχονται τι κριτικέ μα. Αλλά αν δεν υπάρχει κριτική, δεν θα υπάρχει και εμπιστοσύνη. Τα λάθη μειώνονται, όντω, και η εκτέλεση και η αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης αυξάνεται. Οι υπηρεσίες κάνουν όλο και περισσότερες προσπάθειες για να βελτιώσουν το σύστημα ελέγχου τους. Βεβαίω, έγιναν κάποια λάθη, τα οποία τα διαπίστωσαν τα άλλα θεσμικά όργανα. Το καλό νέο είναι ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα λάθη. Ε, υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη ΣΕΠΟΛ, το, την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αστυνομία. Ε, τα προβλήματα αυτά οφείλονται σε διάφορους λόγους. Υπάρχουν προβλήματα στα λογιστικά. Ε, υπάρχει πρόβλημα με τη χώρα που φιλοξενεί την, την Ακαδημία. Υπάρχουν προβλήματα με τις, με τους, με τις προκηρύξεις υποβολής ενδιαφέροντος. Υπάρχουν βελτιώσεις από χρόνο σε χρόνο. Ήδη είναι απτά τα, απτές οι βελτιώσεις, παρόλα αυτά τα προβλήματα παραμένουν. Θα ήθελα να προτείνω να αναβάλουμε την απαλλαγή για τον προπολογισμό 2008 της ΕΠΟΛ, της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, όσο δεν έχουν βελτιωθεί οι παρατυπίες. Οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας μας είπαν ότι οι βελτιώσεις θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Σε ό,τι αφορά τους υπευθύνους αυτής της Ακαδημίας, μας υποσχέθηκαν, όπως σας είπα, να κάνουν ό,τι μπορούν, να κάνουν το δύναμη. Σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλεγχο στις διάφορες υπηρεσίες, Μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και πώ. Μπορούμε καταρχά να συνεχίσουμε τι προσπάθειε, ούτω ώστε να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία. Μπορούμε να προωθήσουμε μέτρα απλούστευση των κανόνων των λογιστικών. Και τρίτον, να εξετάσουμε μια πρόταση που έκανε το ελεκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά την καλή λειτουργία αυτών των υπηρεσιών. Ευχαριστώ κύριε Κάλφα. Κύριος Πίπερ για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, θέλω να κάνω μερικέ ε, παρατηρήσει σε σχέση με τη διαδικασία διεύρυνση και την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Υπάρχει η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τα κονδύλια προ την Τουρκία. Εμεί είμαστε απογοητευμένοι από αυτά τα οποία αναφέρει το Ελεκτικό Συνέδριο, διότι δηλαδή τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν από την Κομισιόν χωρί καμία στρατηγική και χωρί καμία αξιολόγηση τη αποτελεσματικότητό του ήδη με το, νέο, με το εργαλείο, νέο εργαλείο ΙΠΑ από το 2007 ήταν απαραίτητο να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών των χρημάτων και πρόκειται για 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να ξέρουμε τώρα πότε θα υπάρξει μια πραγματική δυνατότητα πολιτικού ελέγχου σε σχέση με την αξιολόγηση αυτών των κονδυλίων. Το, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ζητεί λοιπόν από την Κομισιόν να κάνει μια μεταρρύθμιση του προγράμματος ΕΠΑ ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μια, μια αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών χωρίς αυτή την αξιολόγηση θα πρέπει να παγώσουν αυτά τα κονδύλια στο επίπεδο του 2006. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια ευελιξία για αυτό το εργαλείο προενταξιακής βοήθειας και προς τις χώρες της ε, γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε λοιπόν να θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρί να αποδίδουν καρπού. Ο στόχο μα είναι δεν είναι να αναμειχθούμε στα θέματα τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε να δακτυλοδεικτήσουμε ειδικά την Τουρκία. Απλώ θεωρούμε ότι όταν πρόκειται για δημόσια κονδύλια είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδρούμε σε περιπτώσει κακοδιαχείριση. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια εξαίρεση για την Τουρκία. Εάν έχουμε μια τέτοια στάση, δεν θα μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ούτε στην Κροατία, ούτε στη Ρουμανία, ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε άλλες χώρες. Γι' αυτό ζητώ από την Κομισιόν να δώσει μια καλύτερη πολιτική κατεύθυνση ώστε να υποστηριχθεί πράγματι η προενταξιακή πορεία της Τουρκίας με τρόπο ο οποίος βοηθάει την τουρκική κοινωνία. Ευχαριστώ κύριε Πίπερ. Σάλτε μου για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και για τη σχετική έκθεση. Νομίζω ότι την έχουμε μπροστά μας αυτή την έκθεση. Είναι η πιο επικριτική από όλες τις εκθέσεις που μας δώσατε προς εξέταση. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ε, είναι ασύνηθες ένα θεσμικό όργανο να δώσει απαλλαγή στον εαυτό του εφόσον το κάνουμε θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο ανοιχτοί, ακόμη πιο υπεύθυνοι. Αυτή η έκθεση μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αυτοελεγχθούμε με τρόπο σωστό. Ε, καλά τα πάμε, δεν λέω, αλλά νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις επικρίσεις για να βελτιωθούμε θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθεί τις εργασίες μας. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στο, στην ιστοσελίδα μας και στις εκθέσεις μας. Θα πρέπει να έχει επίσης πρόσβαση στις επικριτικές εκθέσεις. Θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλους τους τομείς ο πολίτης και στους επικίνδυνους, ευαίσθητους τομείς. Επίσης, ο τρόπος διαχείρισης θα μπορούσε να βελτιωθεί, θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο διαφανής και για μας και για τους πολίτες, ούτω ώστε να καταλαβαίνουμε όλοι πώς οργανώνεται ο έλεγχος. Μοιάζει εύκολο να το λέει κανεί, αλλά δύσκολο να το κάνει. Δεν έχει νόημα να ξεδεύουμε χρήματα για να βελτιώνουμε τα γραφεία μας, ας πούμε. Κανονικά θα πρέπει να έχουμε μόνο μία έδρα. Έλεγχος διαχείριση καταρχήν και έλεγχος για τα λεφτά των φορολογούμενων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτές οι αρχές θα πρέπει να ισχύουν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη σε αυτή την έκθεση πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση, ε, ασκούμε αυτοκριτική και αυτό θα μας κάνει και πιο αξιόπιστος όταν ασκούμε κριτική σε άλλους. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ακούστηκαν πολλά πράγματα, γι' αυτό θα περιοριστώ σε δύο. Καταρχά για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου. Αν θέλουμε να ελέγξουμε του άλλου, θα πρέπει να είμαστε και αυτοκριτικοί. Και ο κύριο Στά νομίζω ότι παρουσίασε μία έκθεση α, την οποία μπορώ να υπερψηφίσω, θα μπορούσα να είχα υπερψηφίσει πριν από 6-7 ή 7 χρόνια α, πολύ πρό, πρόθυμα. Αλλά μέσα σε αυτά τα 6-7 χρόνια άλλαξαν πολλά πράγματα, βελτιώθηκαν πολλά πράγματα η επιστροφή των ταξιδιωτικών ε, εξόδων με βάση τα πραγματικά έξοδα του καθενός. Αυτό που είναι κρίμα είναι ότι όλες αυτές οι βελτιώσεις δεν αναφέρονται όλες στην έκθεσή του. Και ελπίζω μέχρι την ψηφοφορία να διορθώσει την έκθεση, ούτως ώστε να γίνει πιο ισορροπημένη το κείμενό του. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, μια γενική παρατήρηση. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε μία συζήτηση, ε, δύσκολη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Γιατί έχουμε και νέες ε, αρμοδιότητες, νέα καθήκοντα μετά την υιοθέτηση τη συνθήκης της Λισαβόνας. Επομένως θα έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα να κάνουμε. Θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και κατά συνέπεια θα πρέπει και το ελεκτικό συνέδριο να μπορεί να ελέγχει τα πράγματα. Δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην επαλήθευση των λογαριασμών. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπορεί να ελέγξει ουσιαστικά έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Απλώ επαληθεύει. Αν θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα προπολογισμό ο οποίο να διέπεται από έλεγχο, θα πρέπει το ελεγκτικό συνέδριο να λειτουργεί όλο διόλου διαφορετικά. Νομίζω ότι στο μέλλον, όταν κάνουμε τέτοιε συζητήσει για το προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να είναι παρόν. Να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ σκοπεύει να ρυθμίσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ την κυρία Ντελάνιε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Βόν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να μιλήσω για την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή εργασία την οποία έκανε μαζί πολλούς άλλους. Θα ήθελα να σας πω ότι βελτιώνουμε την διαφάνεια και την απόδοση των χρημάτων των καταναλωτών. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν βελτιώσεις και γι' αυτό δεν ε, είμαι βέβαιος ότι όλες οι συστάσεις ε, είναι βελτιωτικές. Παραδείγματος χάρη οι βελτιώσεις ε, του κτηρίου αυτού που θα είναι πολύ δαπανηρές. Επίσης η αύξηση του στόλου αυτοκινήτων του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ήδη περιλαμβάνονται ή στις προτάσεις για το 2011 παραδείγματο χάρη την τηλεόραση Europal TV και την έκκληση για να υπάρχει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική ε, κτηρίων η οποία να μας βοηθήσει στο μέλλον. Θα έπρεπε λοιπόν να καλύψουμε και τα θέματα τα οποία έχουν ε, ήδη ε, ολοκληρωθεί. Έχουμε όμως και θετικά παρατηρήσεις τις οποίες θέλουμε να στηρίξουμε παραδείγματο χάρη την ε, μείωση ε, των ε, γραφών θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη μείωση βλέπουμε τα βουνά το, της χαρτούρας η οποία τυπώνεται καθημερινά. Θα έπρεπε λοιπόν να αποφύγουμε επίσης τις επικαλύψεις να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και θα υπάρξουν και νέες τροπολογίες για τον τροπολογισμό του Κοινοβουλίου του 2011 διαχείριση του κινδύνου. Επίση είναι ένα θέμα που χρήση βελτιώσεω, αλλά γενικώ πιστεύω ότι έχουμε μία ισοσκελισμένη συζήτηση. Θα υπάρξει απαλλαγή για τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ελπίζω ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θα συνεχίσει να εξασκεί υπεύθυνα τι ε, αρμοδιότητέ σου και να προτείνει βελτιώσει όσον αφορά το σύστημα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ρούμπικ για δύο λεφτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι χάρηκα διότι αυτή την εβδομάδα χρειάστηκε να έρθω απλώς στο Στρασβούργο και όχι στις Βρυξέλλες που είναι πιο κοντά στο σπίτι μου και παρόλες τις διαταραγμένες αεροπορικές μεταφορές μπόρεσα να φτάσω απρόσκοπτα. Όσον αφορά την ε, εργασία της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, για αυτή την εβδομάδα έχουμε ένα μεγάλο πακέτο σαν αυτό που κρατώ, που μας δείχνει τι έχουμε να διεκπαιρεώσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να είχαμε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, να μπορούμε να τα παρακολουθούμε ηλεκτρονικά ε, και να έχουμε μπροστά μας στη γλώσσα μας για την ψηφοφορία, την τροπολογία στη γλώσσα μας για να γίνεται απρόσκοπτα η ψηφοφορία. Διότι οι ψηφοφορία είναι το μεσημέρι και καλό θα ήταν να μην χρειάζεται να κουβαλάμε όλα αυτά τα τεράστια ε, χαρτοβασίλια και να μπορούμε να έχουμε υπολογιστές και να είμαστε ενήμεροι τεχνολογικά. Τώρα, ε, αν δούμε ε, πόσο έχει αυξηθεί η γραφειοκρατία ε, θεωρούμε ότι αυτό προκαλεί μεγαλύτερες δαπάνες για όλους και για την διαχείριση και για τη διοίκηση και γι' αυτό θα έπρεπε να καταρτήσουμε μία ομάδα εργασίας η οποία θα πρέπει να αφιερωθεί στο σωστό υπολογισμό και να μειώσει τη γραφειοκρατία κατά 25% και όχι αυτό που έγινε ε, τους τελευταίους μήνες όπου αυξήθηκε η γραφειοκρατία κατά 50%. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει, διότι έχουμε πολλές χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση και αν ε, το Περιφερειακό Ταμείο μπορεί ε, να προβεί ε, σε πρόβλεψη επενδύσεων και όχι απλώς καταναλωτικές πιστώσεις και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ λογικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ. Και ε, η, τέλος η κυρία Τικάου για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, Επίτροπε. Θα ήθελα <clears throat> να αναφερθώ στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2008 και συγκεκριμένα αναφέρομαι στον προϋπολογισμό της Κομισιόν και των αποκεντρωμένων φορέων. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της ε, Δανίας, των κάτω χωρών και άλλων χωρών που θελήσαν να προβούν σε εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Πιστεύουμε ότι αν ακολουθήσουν και οι άλλες χώρες το παράδειγμά τους, θα προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση σημαντικών προόδων. Ζητούμε λοιπόν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει συστάσεις σε σχέση με την εκπόνηση εθνικών δηλώσεων σε σχέση με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ερευνητικά προγράμματα, πιστεύω ότι οι τωρινοί πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μια έρευνα άξια του ονόματός της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να προκύψουν σημαντικές βελτιώσεις για το μελλοντικό πρόγραμμα, ερευ... πρόγραμμα πλαίσιο στον ερευνητικό τομέα. Αναφέρομαι επιπλέον και στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Φορέα για τον έλεγχο των δεδομένων. Μέσα στον ισολογισμό αυτού του φορέα υπήρχαν έσοδα 143 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο φορέας αυτός έχει μπορέσει να συλλέξει σημαντικού πόρους σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ω εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος όχι μονάχα και ο έλεγχο των κονδυλίων που αφορούν τι άμεσε ανάγκε αυτών των φορέων, αλλά να δούμε πώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι άλλοι πόροι που προέρχονται από αυτό το φορέα μετά το 2012. Ερχόμαστε στη διαδικασία κάστη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμεί θέλουμε να είμαστε μια ένωση που θα, την δεχόν, τη δέχονται οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό και κεντρικό να ξέρουν οι πολίτε τι κάνουμε με τα χρήματα των φορολογουμένων. Αυτή ήταν και η έτσι της κυρίας Σάλτε Μούσε, να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και επομένως εδώ είναι κάτι από το οποίο θα δοκιμαστεί και θα κριθεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει και μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν οι πολίτες μα τη δυνατότητα να κατανοούν τι σημαίνουν τα έγγραφα της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι στο επίπεδο αυτό να ζητήσουμε από την Κομισιόν να εκπονεί τα έγγραφά της, ιδίως τα δημοσιονομικά και αυτά που έχουμε τον προϋπολογισμό, σε επίπεδο αναγνώσιμο και εύληπτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι πολίτες πόσο μικρός ή πόσο μεγάλος μπορεί να είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτά τα οποία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν μπορούν να ζητούν κάτι όταν δεν υπάρχουν κονδύλια για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να καταλάβουν λοιπόν τα πολιτικά προγράμματα και ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα μπορέσει να προχωρήσει και προς την κατεύθυνση αυτή στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Ζέμπερ. Ο κύριος Μάιερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να κατακρίνω τον οργανισμό βοήθειας προς την Τουρκία το οποίο οπισθοδρομεί περισσότερο από ό,τι να προχωρά και διαπιστώνονται σημαντικά προβλήματα οι πόροι δεν χρησιμοποιούνται σωστά ε, και ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους και τους εξηγήσουμε τι έγινε με τα 800 εκατομμύρια βοήθεια προς την Τουρκία διότι από το 2000 έχουν οι χορηγήσεις τριπλασίαση παρόλο που προσπαθούμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία και επίσης με ενδιαφέρει τι έχει γίνει με την ε, παρακολούθηση των ναρκωτικών διότι στην Τσεχία έχουν ε, ε, νομιμοποιηθεί τα ναρκωτικά από τις αρχές του έτους και έχει δημιουργηθεί ένας τουρισμός υπέρ των ναρκωτικών στη χώρα αυτή. Ο κύριος Κασπάρη τώρα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ε, κύριοι, και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην προενταξιακή βοήθεια, διότι το ελεκτικό συνέδριο λέγει ότι βάσει των ισιών των προγραμμάτων δεν είναι σε, σε θέση να αποδείξει ότι οι πόροι έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες που δεν μπορούν να ελεγχθούν και η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού εξέφρασε σαφώς τη θέση του ε, την ε, ε, γνωμοδότηση και τώρα υπάρχει ισχυρό λόμπι από την Τουρκία. Το θέμα δεν δεν, που μας απασχολεί δεν είναι αν θα προσχωρήσει η Τουρκία ή όχι, αλλά αυτό που πρέπει να ελέγξουμε είναι αν τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά, αν οι πόροι καταλήγουν σε αυτούς οι οποίοι είναι οι σωστοί αποδέκτες και ε, εάν προχωρούμε σωστά. Δηλαδή, θα ήθελα λοιπόν παρακαλώ ε, να, να λάβετε τη σωστή απόφαση όταν τελικά θα ψηφίσουμε του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κασπάρη. Ο κύριος Γκόνς. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, Εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο είναι αντίθετο στη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε θα απορρίψουμε την απαλλαγή ασχέτως των πιστηρίων θα μπορούσαμε να απορρίψουμε την οποιαδήποτε μελλοντική, ε, μελλοντική δαπάνη και να αποδεχθούμε την απαλλαγή ε, του παρελθόντος εάν είχαμε επαρκή πιστήρια αλλά δεν θα δεχθούμε την απαλλαγή διότι υπάρχουν πολλές αταξίες δεν αμφισβητούμε ε, την την σωστή χρήση ε, αρκεί να ε, αιτιολογηθεί ο στόχος. Θα πάρουμε μια κριτική αντιμετώπιση για όλα τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Γκρόνς και θα καταλήξουμε με την κυρία Γκλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την απαλλαγή. Η Απαλλαγή του προπολογισμού του 2010 είναι πάντοτε μια ευκαιρία για προβλέψεις και ε, ιδίως προβλέψη χρειάζεται ε, για όλους αυτούς τους οργανισμούς που έχουμε καταρτήσει οι οποίοι θα πρέπει να επανδρωθούν με τις ε, οικονομικές δυνατότητες και ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούν να εργαστούν. Αναφέρομαι εις τον οργανισμό που είναι υπεύθυνο για την χημεία και θα περιλάβει στο μέλλον και τα διοξίδια. Θα πρέπει λοιπόν ε, στο μέλλον να είναι αποτελεσματικός ο οργανισμός αυτό στην εργασία του και θα παρακαλούσα να στηρίξουμε αυτό τον οργανισμό για να μπορέσει στο μέλλον να εργαστεί αποτελεσματικά προς όφελός μας. Ευχαριστώ την κυρία Κλάς. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Σεμέτα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω ξανά ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη για να σημειωθεί, σημειωθεί περαιτέρω πρόεδρο, πρόοδος για να βελτιωθεί η ποιότητα των εξόδων. Ε, θα κοιτάξω προσεκτικά τις αποφάσεις απαλλαγής που θα υιοθετήσει το Κοινοβούλιο σε δύο εβδομάδες και η Κομισιόν θα εξασφαλίσει το σωστό follow-up, τη σωστή συνέχεια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίσης για την πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση Ακούστηκαν πολλές ιδέες, ενδιαφέρουσες ιδέες και θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες από αυτές. Καταρχάς, την εθνική διαχείριση και τις εθνικές δηλώσεις. Ο κ. Στάς έθεσε αυτό το θέμα και άλλοι βουλευτές. Θα ήθελα να σε υπενθυμίσω ότι μαζί με τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι στείλαμε μια επιστολή στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού που λέει ότι στην επερχόμενη μεταρρύθμιση του κανονισμού θα αναθεωρήσουμε το θέμα που αφορά τις δηλώσεις, θα κάνουμε προτάσεις για απλούστευση, θα εισάγουμε την έννοια του επιτρεπόμενου ορίου σφάλματος. Ο κύριος Σόντεγκαρτ μίλησε, μίλησε ιδίω για τα διαφθορτικά ταμεία. Ε, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου τέθηκε από την κυρία Χέρτσοκ. Συμφωνώ με τις απόψεις της. Την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε στα πλαίσια της στρατηγικής ε, για το 2012 ε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σκεφτούμε αυτά που είπε ο κ. Σοντή και κάποιοι άλλοι βουλευτές για τη διαδικασία της απαλλαγής. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το πώς θα βελτιώσουμε τη διαδικασία της απαλλαγής για να αλλάξουμε αυτή τη διαδικασία και με το συντομότερο δυνατόν. Το συντομότερο δυνατόν. Ε, κοιτάξτε, σήμερα έχουμε φτάσει το 2010. Συζητάμε ακόμα την απαλλαγή του 2008. Άρα τι αλλαγέ θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει για το 2009. Θα πρέπει να γίνει μια ευρεία συζήτηση με το ελεκτικό συνέδριο, όλους τους ενδιαφερόμενους. Ε, συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις του κυρίου Ντί, λοιπόν, για το θέμα αυτό της αλλαγής και της επιτάχυνσης της διαδικασίας. Επίσης, το θέμα της αποτελεσματικότητας και της ορθής δαπάνης των κοινοτικών κονδυλίων. Στην ε, Γενική Στρατηγική Ελέγχου θα εστιάσουμε στον τρόπο βελτίωσης του ελέγχου. Θα συμπεριλάβουμε και το θέμα της ε, αποτελεσματικότητας στον τρόπο που δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για το θέμα της Τουρκίας. Ακούστηκαν συστάσεις για να βελτιωθούν οι στόχοι και η παρακολούθηση της πρόοδου. Θα το εξετάσουμε. Θα πρέπει σε όλους τους τομείς να βελτιώσουμε την ποιότητα των δαπανών. Από τους στόχους μέχρι την μελέτη αντικτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί για να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτή η πρόοδος είναι αποτέλεσμα και της δικής σας δράσης ως ε, οργάνου αρμόδιου για την απαλλαγή. Όπου δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, ε, είσαστε πάντα επικριτικοί, αλλά είσαστε υποστηρικτικοί εκεί όπου σημειώνεται πρόοδος. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θα πρέπει να περάσει στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν να καταλήξω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια καλύτερη οικονομική διαχείριση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ευχαριστούμε κύριε Σεμέτ. Τώρα Τώρα έχουν τη δυνατότητα οι συγητέ να δευτερολογήσουν και δίνω πρώτα το λόγο στον κύριο Γκάιγερ. Για να γραφεί σωστά στα πρακτικά, εκπροσωπώ τον εισηγητή και όπως και πολλοί άλλοι αυτή την εβδομάδα ήταν θύμα των ε, προβλημάτων ε, συγκοινωνιών αλλά ευχαρίστω τον αντιπροσωπώ και θα μπορέσω να κάνω και ε, ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά τη συζήτηση. Καταρχήν Αξιότιμη κύριε Επίτροπε Σεμέτα, Προς μεγάλη μου ικανοποίηση σημειώσατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει διαβήματα κατά τρόπον ώστε να απολογηθούν οι και να ε, ενισχυθούν ε, τα μέσα ελέγχου των ε, διοικήσεων, δηλαδή τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που διαχειρίζονται ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κινούνται σωστά διότι ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των λαθών που γίνονται στη διαχείριση των πιστώσεων οφείλονται στα κράτη-μέλη. Οπότε ε, θα, δεν είμαι ε, ικανοποιημένος όταν ακούω τους ε, Ευρωπαίους συντηρητικούς και τον κύριο Σαρνέσκι ότι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, και κατακρίνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, τις ε, και λέγουν ότι δεν θα τις ε, χορηγήσουν απαλλαγή. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να εγκαλέσει κανείς και τα κράτη-μέλη και τις, τις εθνικές διοικήσεις οι οποίες πρέπει να συνεργάζονται σωστά και έτσι δεν είναι σωστό όταν οι εκπρόσωποι του συντηρητικού κόμματος έρχονται και προσάπτουν ευθύνες οι οποίες ανήκουν σε άλλους. Θα ήθελα όμως εδώ να σας πω ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού υπερψήφισε την έκθεση με μικρή πλειοψηφία και σε τέτοιο σημείο ώστε ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου προσπάθησε ε, να, ε, να εξηγήσει στον εισηγητή ότι εδώ εξι, ε, αναφερόμασταν στην συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι της Τουρκίας διότι εδώ δεν πρόκειτο μόνο για χρήση χρημάτων χρημάτων το φορολογούμενο, αλλά πού πηγαίνει η ε, αναπτυξιακή βοήθεια για την Τουρκία η προενταξιακή βοήθεια για την Τουρκία και πιστεύω ότι το, η απαλλαγή του προπολογισμού δεν είναι το σωστό σημείο για να παρουσιαστεί αυτό. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Σεμέτα και τι υπηρεσίε τη Κομισιόν για τα θέματα τη ανθρωπιστική βοήθεια, τα οποία έδειξαν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί μου. Θέλω να εκφράσω επίση την αναγνώρισή μου και την ευγνωμοσύνη μου στην Ισπανική Προεδρία για τι προσπάθειε που έκανε στα πλαίσια τη διαδικασία απαλλαγή για να προβεί τη διαθεσιμότητά τη να προβεί σε μια συζήτηση για μια νέα διαθεσμική συμφωνία για τα θέματα αυτά. Θέλω επίση όμω να αναφέρω και την απόρριψή μου λόγω της αυτοσχέδιας αυτής διαδικασίας που δεν κάλεσε επίσημα ούτε το ελεκτικό συνέδριο ούτε το Συμβούλιο με τις 9 το πρωί τουλάχιστον. Θέλω επίσης να επικρίνω την ε, απουσία αυτή που δεν δίνει το πρέπον κύρος στην συνεδρίαση αυτή και στον έλεγχό μας. Εάν θέλουμε να αναλάβουμε πραγματικά τις ευθύνες μας, τις νέες ευθύνες, θα πρέπει να έχουμε όχι οπορτουνιστική, αλλά εμπεριστατωμένη έρευνα των στοιχείων του προπολογισμού και τη απαλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου μου και ιδίω την κυρία Χόλμαϊερ για τη συνεργασία τη και όλοι οι συνάδελφοι που μπορέσαν να εξασφαλίσουν μια μεγαλύτερη ε, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στον έλεγχο τη αναπτυξιακή βοήθεια. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι οι πολίτε θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την αναπτυξιακή βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούν να υπάρχει μια μεγαλύτερη έκταση και ορατότητα αυτή τη βοήθεια. Εμά όμω μα απασχολεί γιατί υποστηρίζουμε κάποιε κυβερνήσει μέσω άμεσου άμεση υποστήριξη στον προπολογισμό τη χωρί να υπάρχει αυστηρό έλεγχο, ιδίω όταν πρόκειται για περιπτώσει σκανδάλων διαφθορά, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράξη κοπημάτων, όπω 21 Απριλίου κτλ. Οι σημαντικέ αυτέ πρόοδοι λοιπόν που έχουμε διαπιστώσει σημαίνουν ότι εμεί θα πρέπει να εγκρίνουμε και το 7ο, 8ο και 9ο έτα. Ταμείο Αλλά ζητούμε να υπάρξουν και περαιτέρω βελτιώσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει ότι το νέο διαθεσμικό πλαίσιο που θα δημιουργηθεί μετά από την Λισαβόνα να μην ανατρέψει τι ε, επιτυχίε που έχουμε επιτύχει, ώστε οι πολίτε μα να εξακολουθούν να είναι περήφανοι για την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγιάλα. Ακολουθεί ο κύριο Στάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που αντέδρασαν στην έκθεσή μου και θα ήθελα όλος ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον κύριο Ήταλα, τον κύριο Γκάγιαρ, την κυρία Σάντε Μόζερ, την κυρία Λάγκε και τον κύριο Βόλκερ. Όλα έχουν υποθεί, νομίζω. Αλλά θέλω να εκφράσω την έκπληξή μου σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτής της, την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Δεν ε, είμαι για πρώτη φορά εισηγητής σε τέτοια έκθεση για απαλλαγή ε, και βλέπω ότι υπάρχει, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ε, την πρώτη και δεύτερη φορά ήταν εύκολες οι κριτικές, αλλά την τρίτη φορά ε, έχω την αίσθηση ότι οι επικρίσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια έλλειψη αυτοκριτικής. Κάποιοι συνάδελφοι ε, μου επιτέθηκαν στον, στον τύπο και μου είπαν ότι με αυτά που γράφετε ουσιαστικά δίνεται τροφή ε, στους επικριτές μας. Εγώ είμαι και φιλοευρωπαϊστής, αλλά ξέρω να κάνω και αυτή, αυτοκριτική. Και νομίζω ότι όταν νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να βελτιωθούν, το λέω. Παραδείγματο χάρη για αυτό το Ταμείο Συντάξεων, το Εθελοντικό Ταμείο Συντάξεων. Ε, έχω αρνητικά πράγματα να πω και όταν πιστεύω κάτι τέτοιο και έχω κάτι να πω, το λέω. Συχνά οι ευρωσκεπτικιστές τρέφονται από τις μισοαλήθειες και τα μισοψέματα. Γι' αυτό πρέπει να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Δεν θα αλλάξω κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει στην έκθεσή μου. Αυτή είναι η η θέση μου. Ο κύριος Τσαρνέκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέιερ, ο οποίος ανέφερε ότι μερικές φορές λέω τις πραγματικές μου σκέψεις. Κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακό το πώς φέρεται το Συμβούλιο. Ε, όταν ξεκίνησα την ομιλία μου ε, δεν ήταν εδώ και τώρα πάλι εξαφανιστεί. Όταν είναι να ακούσει κριτική, εξαφανίζεται το Συμβούλιο. Έχω κάνει εκθέσεις για 7 ε, κοινοτικά όργανα, κοινοτικά θεσμικά όργανα. Για τα έξι, τα πράγματα λίγο πολύ ήταν καλά. Αλλά υπάρχει ένα για το οποίο υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και παρατυπίες. Πέρσι ήταν έτσι. Και το ίδιο είναι και φέτος. Δεν θέλω όμως να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου τα έγγραφα που θα λαμβάνουμε θα αφορούν το 2008, αλλά το 2007. Τόσο θα έχουμε καθυστερήσει. Ε, υπάρχει πρόβλημα με την έλλειψη τάξης ε, στο εσωτερικό του Συμβουλίου. Όλοι είναι ισότιμοι, όλα τα όργανα είναι ισότιμα, αλλά το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι πιο πάνω από τους ίσους. Όπως τη φάρμα των ζώων του Όργουελ. Κάποια ζώα πιστεύουν ότι είναι παραπάνω από τα υπόλοιπα. Το Συμβούλιο είπε ότι μπορεί να δεχθεί να σταματήσει αυτή η Συμφωνία Κυρίων του 1970. Ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου αναγνώρισε παρόλα αυτά ότι τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι και εκλεγμένο άμεσα από τους πολίτες. Ευχαριστώ. Κυρία Ματιέου, για να κλείσουμε την πρώην μας ε, συνεδρίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές αφενός που συνεργάστηκαν μαζί μου για την εκπόνηση των, ε, της έκθεσής μου και τη γραμματεία της Κομισιόν γιατί ήταν δύσκολη η έκθεση και χρειάστηκε της Επιτροπής μάλλον Προελέκτου Προϋπολογισμού για την υποστήριξη που μου έδωσαν και θέλω να πω ότι συμμετέχω στις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από όλους τους συναδέλφους, ιδίως αυτές που έχουν να κάνουν με τη μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των κοινωτικών κονδύλιων, κάτι το οποίο είναι απόλυτα θεμητό. Θα ήθελα να υπενθυμίσω εν κατακλείδη ότι οι αποκεντρωμένοι φόροι για τους οποίους αναφερθήκαμε έχουν και ένα πολιτικό έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσω αυτό και αυτή η πολιτική ευθύνη τους είναι σημαντική. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο υπόκεινται αυτοί οι φορείς και το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε σύμπνια με το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος των αποκεντρωμένων φορέων από τα τρία θεσμικά μας όργανα. Ορισμένοι από τις αποκεντρωμένες φορείς εκτελούν πράγματι το πρόγραμμά τους, άλλοι φορείς δεν είναι τόσο ευήκοοι και το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν όροι περιοριστικοί από τη δική μας πλευρά και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε καλύτερα στο μέλλον για το πώς θα γίνει το έργο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία ματιού. Θέλω να σας υπενθυμίσω βλέποντας τα πρακτικά τώρα της προηγούμενης θητείας το Συμβούλιο έλαβε μονάχα μία φορά θέση και παρέστη σε μια τέτοια διαδικασία στο επίπεδο της δεύτερης ανάγνωσης και λόγω αυτό, αυτού ανεβλήθη πέρσι η, η διαδικασία απαλλαγή. Επομένω, δεν είναι σωστό ότι το Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να παρισταθεί. Εν πάση περιπτώσει, κλείνει η συνεδρίαση και θα ξεκινήσουμε και πάλι στι 3 ώρα το απόγευμα.